Ε, παρακαλώ να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Θα περιοριστούμε μόνο στο ένα θέμα, ε, στο negotiations on the MFF ε, lessons to be learned and the way forward. Έχουμε εισηγητή τον κύριο Γιάνν Όλμπριχτ. Διαπραγματεύσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Διδάγματα που πρέπει να, να αντιληφθούν και μελλοντικέ προοπτικέ. Ο κύριο Όλμπριχτ. Θα μιλήσω πολωνικά, πρόεδρε. Ε, Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε ένα σχέδιο γνωμοδότησης για μια έκθεση πρωτοβουλίας την οποία προετοιμάζει η Επιτροπή Προπολογισμών. Η έκθεση λοιπόν αυτή της Επιτροπής Προπολογισμών έχει να κάνει με τα διδάγματα τα οποία πρέπει να αντληθούν και τις μελλοντικέ προπτικές από τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η γνωμοδότησή μου, το σχέδιο γνωμοδότησης είναι αρκετά σύντομο όπως το βλέπετε και επικεντρώνονται σε κάποια ενδιαφέροντα σημεία σε σχέση με τις διαπραγματεύσει για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε εντοπίσει. Πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να αποφύγουμε να επαναλάβουμε στο μέλλον κάποια από τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, ακολουθώντας βέβαια πάντα τις διατάξεις ε, της συνθήκης. Προβλέπεται μία αποκλειστική διαδικασία συμφωνίας, σύμφωνης γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με ένα κείμενο το οποίο υποβάλλει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ως προς αυτό εμείς κάνουμε τις εξής προτάσεις. Υποβάλλουμε μάλλον μια πρώτη δική μας πρόταση και στη συνέχεια τον Ιούλιο μια δεύτερη σχετική πρόταση και στη συνέχεια προβλέπεται μια συζήτηση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι τα όσα πρότεινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των πραγματεύσεων δεν ανταποκρίνονταν στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δική μου λοιπόν γνωμοδότηση βασίζεται στα εξή. Θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν ουσιαστικά δύο διαδικασίες. Πρώτον, η διαδικασία της προετοιμασίας των δημοσιονομικών προοπτικών και από την άλλη μια διαδικασία για την προετοιμασία της νομικής βάσης για τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της ε, περίοδου προγραμματισμού. Στη γνωμοδότησή μου λοιπόν εξηγώ σαφέστατα ότι οι δύο αυτές διαδικασίες πρέπει από νομικής πλευράς να είναι απόλυτα χωριστές. Δηλαδή θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις συζητήσεις για το πολιτές νομικό πλαίσιο και τις συζητήσεις για τη μία μόνο νομική βάση για τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, το Ταμείο Συνοχής. Το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει και αυτό να το αξιολογήσουμε, να το αναλύσουμε και θα πρέπει να δούμε αν τελικά η πολιτική συνοχής όντως ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη. Ένα σημαντικό σημείο της γνωμοδότησής μου είναι το ακόλουθο. Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την περίοδο τι ακριβώ επιπτώσει έχουν τελικά στον κοινοτικό προπολογισμό. Αναφέρθηκε στα ζητήματα αυτά και ο Γενικό Ευθυντή κ. Ντεφά σήμερα το πρωί. Μέχρι τα τέλη του έτου πρέπει να δούμε αν τελικά έχουμε του απαραίτητου πόρου για να καλύψουμε τι ε, δαπάνε που έχουμε αναλάβει και αν έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε στη συνέχεια με ένα απόθυμα το οποίο θα έχουμε και τα επόμενα έτη τα οποία θα ακολουθήσουν σε περίπτωση που οι πόροι δεν είναι αρκετοί. Το πρόβλημα είναι ότι ενδεχομένω να μην καταφέρουμε να καλύψουμε όλα τα αιτήματα πληρωμών των κρατών μελών καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου προγραμματισμού. Πρέπει λοιπόν να δούμε καταρχάς ποιο είναι το καθεστώς της όλης συζήτησης για το Ταμείο Συνοχής και στη συνέχεια θα πρέπει να καταφέρουμε, όπως σας είπα, να διαχωρίσουμε τη συζήτηση αυτή από τη συζήτηση που γίνεται για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο θα λάβουν οι σκιώδεις Ποιος είναι... Ο κύριος Φρανσουά Αλφωσή. Είσαι έτοιμος Φρανσουά. Ε, κύριε Ernst. Εμένα με λένε Κωνσταντσε Κρέλ κύριε Πρόεδρε. Η Κορνέλια Έρνστ είναι από άλλη πολιτική ομάδα. Είναι λίγο γκούε. Εντάξει. Δεν πειράζει, δεν ξέρουν ε, αυτά ο κόσμος. Είμαι σκιώδης συγγήτρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Okay. Δεν το έχουμε εδώ, λέει ο πρόεδρος. Ε, ναι, είμαι, είμαι όμως. Παραμένω ε, ακόμα στη σοσιαλδημοκρατική ομάδα, δεν έχω αλλάξει. Παραμένω, ε, λέγομαι Κωνσταντζε Κλέρ, ούτε όνομα άλλαξα. Και είμαι και σκιώδη συγγήτρια, όλα αυτά μαζί. Όχι, ευχαριστώ, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάνν Όλμπριχτ. Ε, πάρα πολύ γρήγορα δούλεψε και ήμασταν υποχρονική πίεση για την γνωμοδότηση αυτή. Με όλα αυτά που είπε συμφωνώ απολύτως 100%. Πλην όμως έχω ένα πρόβλημα. Εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε επιβάλει στον εαυτό μας αυτό που συναποφασίσαμε στη συναπόφαση και ε, επέμεινε και η Επιτροπή Προπολογισμών να μην αναμειγνύεται με τα υπόλοιπα. Παρόλο που οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων σε συνόδους κορυφής έχουν ε, λάβει κάποιες αποφάσεις εκ των προτέρων που μας ε, δυσκόλεψαν τις διαπραγματεύσεις στους τριμερείς διαλόγους. Εν πάση περιπτώσει, κάτι που δεν γνωρίζω και πώς μπορώ να κάνω τροπολογία σχετικά είναι το εξής. Τι γίνεται με το αποθεματικό των επιδόσεων, διότι εκεί έχουμε τη διαδικασία συναπόφασης και η αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων με τις αποφάσεις που πήρανε και για τα ποσά, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μας έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση που δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε αυτό το αποθεματικό επιδόσεων. Γιατί σε περίπτωση που το αρνούμαστε ε, θα ε, ε, έπρεπε να αναπροσαρμοστεί το δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν ξέρω τελικά πώς θα κανονίσαμε αυτά. Ότι κάποιες οικονομικές αποφάσεις μπορούν να παρακάμπτουν την νομοθεσία ή δεν επιτρέπεται να ε, την επηρεάζουν. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται και πώς μπορούμε να το διατυπώσουμε, γιατί ήταν δική μας απόφαση αυτή. Για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, πρώτα δεχόμαστε τους στόχους και όταν ε, μιλάμε για αναφορές ή διαφορές έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο και όχι με αριθμούς. Και όταν οι αριθμοί δεν ισχύουν και ανατρέπονται, ίσως ανατρέπεται ολόκληρο το πλαίσιο. Δεν ξέρω, ο Γιάν θα μπορούσε να με διαφωτίσει για να το καταλάβω και να το βάλω στις τροπολογίες. Γιατί είναι κονδύλια για την πολιτική συνοχή που έχουν περικοπεί. Αυτό και τίποτα άλλο. Καμία σχέση με αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά. Περιφέρειες που έχουν πολύ καλές επιδόσεις να έχουν τη δυνατότητα η επιπλέον χρηματοδότηση. Όλα αυτά δεν ισχύουν, δεν είναι πια στο αποθεματικό αυτό. Έχουν αναβληθεί όλα αυτά για την περίοδο μετά το 2020. Και νομίζω ότι θα πρέπει να διατρανώσουμε και πάλι και να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ιδρύσαμε ξεχωριστή επιτροπή, όχι μόνο εμείς, το ζήτησαν και άλλες επιτροπές από την αρχή, για να συνεργαστούν πολύ στενά με εκείνους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, με τον προϋπολογισμό, με τα στοιχεία τα αριθμητικά. Καλά κάναμε δηλαδή και ε, συμμετείχαμε από την αρχή σε αυτή την προσπάθεια και στη λήψη των αποφάσεων. Αξίζει να το ξαναγράψουμε στη γνωμοδότηση ότι και την επόμενη φορά θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Αλφονσί. Νομίζω μπορούμε να πούμε ότι επί της ουσίας συμφωνούμε με όσα έχει συντάξει ο κύριος Όλμπρι και με όσα είπε μόλις τώρα η κυρία Κρέλ. Απλώς να θυμίσω τις ανησυχίες μας για τη διάρκεια των δημοσιονομικών ε, δεσμεύσεων στο πλαίσιο αυτού του πολιετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού, ιδίως ό,τι αφορά τη συνοχή. Να θυμίσω στον κύριο Όλμπρικτ ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αναφερθεί και σωστά αναφέρεται στο τρίτο σημείο, στον κατάλογο με τους στόχους, τους πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής συνοχής. Ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόληση, οι δημόσιες επενδύσεις, η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και η Νομίζω ότι θα ήταν καλό να προσθέσετε εδώ την ενεργειακή μετάβαση. Ευχαριστούμε λοιπόν τον εισηγητή για αυτή την έκθεση που μας ικανοποιεί ως ομάδα. Ευχαριστούμε κυρία Άντρε Σμιθ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Όλμπριχτ για την έκθεσή του. Νομίζω ότι ανακεφαλαιώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά τι διαπραγματεύσει του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Θα έπρεπε να είναι πιο εύληπτα τα αποτελέσματα και για τους πολίτες και αυτό είναι μεγάλο μειονέκτημα και βεβαίω βλάπτει τι δημοκρατικέ διαδικασίε που μα ενδιαφέρουν. Δυστυχώ οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων διαπραγματεύονται τη νύχτα κάποιε φορέ σαν να ήταν ε, αράβε έμποροι ο καθένας προσθέτει το δικό του μικρό σκέλος φράσης για να ικανοποιούνται τα διάφορα εθνικά συμφέροντα. Αυτή η μέθοδος διαπραγματεύσεων βλάπτει πιστεύω τη λειτουργία συνολικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποτε όπως οι θεοί του 12 ανακοίνωναν τις μεγάλες τους αποφάσεις ανά τα πρόκειται για δώρο για την ανθρωπότητα, κάπως έτσι φαίνεται να πράττουμε κι εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση ικανοποιώντα εθνικούς εγωισμούς αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου περιορίζεται και από τις εντολές που λαμβάνει κατά τους τρεμερούς διαλόγους. Η πολιτική συνοχής επηρεάζεται από αυτές τις δημοτεύσεις. Καμία τομεακή πολιτική, τις οποίες ε, πρέπει να διαπραγματευτούμε, δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Εθνική Συνεργασία, όπου εγώ παρακολούθησα τις διαπραγματεύσεις από πλευρά της δικής μου πολιτικής ομάδας. Το Συμβούλιο με τι διαδοχικέ προεδρίες δεν έκανε καμία κίνηση. 7% του συνολικού χαρτοφυλακίου της πολιτικής συνοχής έχουμε, που θέλαμε ε, δεν το λάβαμε, αλλά μόνο 2,7%. Και για τα προγράμματα Interreg ε, επιμείναμε πάρα πολύ για να λάβουμε περισσότερα, αλλά το Συμβούλιο αρνήθηκε κατηγορηματικά. Το Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν δεν είχε μεγάλα μέσα πίεση και εδώ να χαιρετήσω το έργο του Προέδρου, της Προέδρου μας, της κυρίας Χιούμπνερ, του κυρίου Φανίστερ Ρόι, του κυρίου Όλμπριχτ και από την Επιτροπή Προπολογισμών του κυρίου Λαμασούρη, οι οποίοι πραγματικά ξεπέρασαν τα όρια όσων μπορούσε να αποσπάσει αυτό το κοινοβούλιο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν έχουμε προγραμματισμό για μια επταετία και το κοινοβούλιο έχει καταφέρει να προστατεύσει κάποιε από τι επενδύσει του μέλλοντο, αλλά το Εράσμου, η βοήθεια προ του πλέον φτωχού, η στήριξη τη έρευνα και τη καινοτομία θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερα κονδύλια στη διάθεσή του. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή λοιπόν να τα προωθήσουμε προωθήσουμε αυτά και να δώσουμε ε, κάθε αξία στο κάθε ευρώ που βγαίνει από τον ε, Ευρωπαϊκό Κορβανά για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει να ξαναδούμε τους πόρους του δημοσιονομικού του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και τα κράτη-μέλη να κάνουν ειλικρινείς προβλέψεις ώστε κάθε φορά να μην βρίσκονται στα χέρια, με έναν ε, πολύ μικρό προπολογισμό στα χέρια τους. Επίσης, για το Ταμείο Λιλεγγύης με ανησυχεί αυτό το κονδύλι που έχει προβλεφθεί. Οι φυσικές καταστροφές ολοένα επαναλαμβάνονται. Με τι πρόσφατες πλημμύρε, το είδαμε αυτό στην Ευρώπη, τι έντονες βροχοπτώσει και τι πλημμύρε. Από ένα δι φτάσαμε στα 500 εκατομμύρια. Μείωση κατά το ίμιση λοιπόν για το ταμείο αυτό, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει και καλύτερη πρόσβαση. Ε, ο αγώνα του ερχόμενου κοινοβουλίου θα είναι να σεβαστεί το Συμβούλιο τη δεσμεύση του, να προβλέψει ιδίου πόρου, ώστε να μην εξαρτώμεθα πλέον μόνο από την καλή βούληση των κρατών μελών και να υπάρχει και μια ενδιάμεση αναθεώρηση ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει έστω και μελλοντικά, να επιβάλλει και τις δικές του πολιτικές επιθυμίες για συγκεκριμένα ζητήματα, κυρίως θέματα όπως αυτό το τομείο της αλληλεγγύης. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς το λόγο, κύριε Φανίστορο. Yeah, Ευχαριστώ πολύ. Είχα διαβάσει το κείμενο, είχα την ευκαιρία ε, προηγουμένως να το δω. Είναι σημαντικό το μήνυμα στο σημείο 4 και 5 ότι θα πρέπει να δούμε στη μετάβαση από τη σημερινή και τη νέα περίοδο πώς θα γίνει αυτή. Με ανησυχεί αυτό. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία και κάποιες δυνατότητες ε, μετάβαση στη νέα περίοδο και μεταφοράς από προηγούμενα αίτια. Αλλά αυτό που είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ανάμεσα στο παλιό και στο νέο έχουμε τεράστιες επικαλύψεις σε λογοριασμούς που δεν έχουν καθαριστεί. Δηλαδή, ήθελα να πω, δεν λέω ότι πήγανε στραβά τα πράγματα ή δεν είναι καλές οι βελτιώσεις, αλλά διαπιστώνω ότι, πώς να το πω, εκκρεμούν ακόμα λογαριασμοί και ξέρουμε περίπου το συνολικό ποσό στον προπολογισμό και το ξέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν έχουν λυθεί αυτά τα θέματα και διανύζονται από χρόνο σε χρόνο. Και ήθελα να το πω αυτό και να το ξέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα με μια καλή λύση που να μπορούμε και εύκολα να την ε, επικοινωνούμε. Ε, έχουν συμφωνήσει για τα οικονομικά στο Συμβούλιο, ε, τα οποία οικονομικά δεν τα ελέγχουν πάρα πολύ λένε Μωρέ, τα ελέγχουν και τα παρελέχουν, αλλά έδειξε μεγάλη επιπολαιότητα το Συμβούλιο με τις υποχρεώσεις. Και τώρα έχουμε τους λογαριασμούς αυτούς που περιμένουν να πληρωθούν. Και ήθελα να το αναφέρω αυτό. Και είναι από τα μεγάλα σημεία τριβής και τα ανισχυτικά που έχουμε και ζούμε αυτό τον καιρό. Εγώ δεν περιμένω τώρα μεταρρύθμιση του συστήματος στη ίμιση της περίοδου Όλοι περιμένουν πλέον την πολιτική το 2018, ας πούμε, το πώληση, για να μπορέσει ε, αυτό να προσαρμοστεί. Δεν κάνω εγώ τέτοια έκκληση. Χρειάζεται περισσότερη εστίαση στα θεματικά και περισσότερη σχέση με τα όσα συμβαίνουν στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες, στα διάφορα προγράμματα και στη συγχρηματοδότηση που χρειάζεται οπωσδήποτε. Εν πάση περιπτώσει δεν ζητώ αναθεώρηση, αλλά ζητώ να λυθεί αυτό το θέμα. Και το λέω και στον εισηγητή, το συντάκτη της γνωμοδότησης. Πρέπει να το διαβιβάσουμε αυτό το μήνυμα και αν τα καταφέρουμε θα είμαι ικανοποιημένος. Ευχαριστώ. Κύριε Όλμπριχτ, θέλετε να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, να απαντήσω στις παρατηρήσεις αυτές. Βλέπουμε καταρχάς ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αναφέρεται βέβαια στην συνθήκη όσον αφορά την εν λόγω διαδικασία, το Ευρωπαϊκό λοιπόν, Συμβούλιο έθεσε την βάση για τις δημοσιονομικές προοπτικές πρώτον αυτών και δεύτερον δημιούργησε μία εντολή διαπραγμάτευσης για το Συμβούλιο Υπουργών. Τελεία και Παύλα, δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα από αυτά. Προετοίμασε αυτή την εντολή διαπραγμάτευσης και στη συνέχεια ακολούθησαν τριμερείς διάλογοι. Εμείς συμμετείχαμε λοιπόν στις διαπραγματεύσεις και εντοπίσαμε εκεί πέρα διάφορα προβλήματα. Η Κωνσταντ Κρέλ είπε πολύ σωστά ότι πρέπει να δούμε ακριβώς σε ποιες επιδόσεις μπορούμε να βασιστούμε. Το είπε αυτό αναφερόμενοι στο αποθεματικό επιδόσεων και πώς αυτό θα, πληρα... θα επηρεάσει τις πληρωμές. Η εντολή λοιπόν αυτή διαπραγματεύσεων θεωρήθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών ως κάτι το περιοριστικό, ως μία υποχρέωση. ενώ για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ πέρα ήταν απλώς μία εντολή διαπραγμάτευσης, η οποία όμως δεν ήταν δεσμευτική ούτε περιοριστική για μας. Οφείλουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στη φάση νη-συν-τρία. 3. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα οι πληρωμές θα αρχίσουν να καταβάλλονται με καθυστέρηση από τη μία χρονιά στην άλλη. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ακριβώς τι λέει σχετικά ο κανονισμός, όπως το είπε πάρα πολύ καλά αυτό και η Κωνσταντ στην παρέμβασή της. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακριβώς όλο αυτό το αρνητικό κλίμα γύρω από τις διαπραγματεύσει, αυτές πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ακριβώς αυτό το αρνητικό κλίμα τελικά οδήγησε στην εντύπωση ότι είχαν ληφθεί κάποιες αποφάσεις ενώ δεν είχαμε καταλήξει τελικά σε συμφωνία. Εμείς δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να θεωρούμε ότι η απλή εντολή διαπραγματεύσεων αποτελεί η λιμένη απόφαση. Πρέπει κάθε φορά να ακολουθούμε τη διαδικασία. Η διαδικασία προβλέπει συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει ήδη λιμένες αποφάσεις. Ακριβώς όμως αυτό χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε πολύ έντονες πολιτικές επιπτώσεις. Αναφερθήκατε στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Όντως, σωστά θέστε το ζήτημα αυτό. Για να απαντήσω και στην κυρία Σάντσες Σμιτ, θα έλεγα ότι ως μέλος της Επιτροπής Προπολογισμών είχα πρόσβαση σε πολύ συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα όσον αφορά την πολιτική συνοχή, δεδομένα που δεν πηγαίνουν σε άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Νομίζω ότι τα αριθμητικά δεδομένα που στέλνει στην Επιτροπή Προπολογισμών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποστέλλονται και στι υπόλοιπε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Συμβουλεύτηκα λοιπόν εγώ αυτά τα δεδομένα, έλαβα γνώση, αλλά νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να συμβαίνει και με τους υπόλοιπους συναδέλφους που συμμετέχουν στις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έθεσε η Μαρή Τερές είναι η δαφική συνεργασία. Εμείς ζητήσαμε ένα ποσοστό 7%, στη συνέχεια υποχωρήσαμε στο 6%. Και σήμερα Αν δούμε πως έχουν τα προγράμματα στην πράξη, βλέπουμε το ποσοστό αυτό είναι ακόμα πιο χαμηλό. Η κατάσταση είναι πραγματικά καταστροφική. Το επιχείρημα το, οποίο προέβαλε το Συμβούλιο ήταν ότι δεν μπορούσαν να αυξήσουν τη συμμετοχή, τα κονδύλια όσον αφορά την εδαφική συνεργασία. Βλέπετε όμως ποιες είναι οι επιπτώσεις. Ίσως αυτό να εξηγεί τελικά και τις πολύ χαμηλές επιδόσεις που έχουμε στην ε, εδαφική συνεργασία. Αλλά αυτό το χρησιμοποίησε το Συμβούλιο σε επιχείρημα για να μην αυξήσει περαιτέρω τα κονδύλια. Ο Λάμπερτ Βανίστε Ρόι αναφέρθηκε στα αιτήματα πληρωμών που δεν καλύπτονται από το... που δεν έχουν πληρωθεί. Ποιος είναι ο αριθμός των πληρωμών που εκκρεμούν ακόμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβα από την ε, Επιτροπή Προϋπολογισμών, βλέπω ότι πάνω από 220 δισεκατομμύρια ακόμα εκκρεμούν, περίπου δηλαδή το 40% των κονδυλίων που προβλέπονται για την περίοδο 2007-2013. 120 δισεκατομμύρια λοιπόν πρέπει να κατανεμηθούν κατά τα δύο ακόλουθα έτη. Και τι θα γίνει όμως με την χρονική περίοδο 2014-2020. Για το έτος 2013 βλέπουμε ότι εκκρεμούν ακόμα κάποια αιτήματα πληρωμών και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει την καταβολή των πληρωμών για το 2014 και τα έτη τα οποία θα ακολουθήσουν. Πρέπει να ρυθμίσουμε, να διευθετήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή πολύ φοβάμαι ότι θα αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικά προβλήματα δεν επιλύσουμε το ζήτημα αυτό. Ε, thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Όλμπριχτ. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι μέχρι αύριο το μεσημέρι, 12 Φεβρουαρίου, διότι πρέπει να ψηφίσουμε στις 24 Φεβρουαρίου και Τώρα θα σταματήσουμε στις 4 και θα ξαναρχίσουμε στις 4 με τις ψηφοφορίες. Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Πριν ψηφίσουμε, έχουμε το σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη, τροποποίηση της απόφασης του ε, Συμβουλίου ε, για την παράταση κατά ένα εξάμεινο από την 1η Ιανουαρίου στις 30 Ιουνίου της ε, ισχύς μειωμένου ποσοστού ε, ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ε, Αζόρα, τη Μαδέρα και τις Ασόρες. Είχα το προνόμιο να είμαι τέλος πάντων ένα αμφισβητούμενο προνόμιο και λόγω ειδικών όρων της συνθήκης αυτές της περιοχές που έπρεπε να υποστούν υπερβολικό κόστος μεταφορών λόγω της απόστασής τους και άλλα πολλά εκτήματα που ίσως ε, παρακολύουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους. Αυτές λοιπόν οι περιφέρειες είχαν ε, ειδική μεταχείριση στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών, μεταξύ των οποίων η μείωση των ειδικών φορών κατανάλωσης. Υπήρξε μια ειδική νομική διαδικασία. Εδώ ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι απλώς συμβουλευτικός. Απλώς γνωμοδοτήσαμε. όπως προβλέπει η διαδικασία για αυτή τη νέα απόφαση του Συμβουλίου. Οι συντονιστές συμφώνησαν ότι δεν έπρεπε να εφαρμόσουμε την απλουστευμένη διαδικασία, δηλαδή το άρθρο 46 του εσωτερικού κανονισμού που μας επιτρέπει δεν επιτρέπει μάλλον να υποβληθούν τροπολογίες, μας επιτρέπει να δράσουμε ταχαίως ε, λέγοντας ναι ή όχι στην ε, πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ρωτήσω λοιπόν εάν συμφωνούν τα μέλη της Επιτροπής να αποδεχτούμε την απλουστευμένη αυτή διαδικασία και εφόσον συμφωνείτε να δώσουμε την καταφατική μας απάντηση στο Συμβούλιο και να αποδεχτούμε το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου. Να σα ενημερώσω παράλληλα ότι αρχικώ η Πορτογαλία είχε ζητήσει πολύ πιο μακροπρόθεσμη παράταση αυτή τη περίοδου, ώστε να προλάβουν να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν και για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα του ειδικού φόρους όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τους νέους κανόνες για την κρατική βοήθεια που θα αρχίσουν να ισχύουν από τον Ιούλιο φέτος. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση είναι να υπάρξει παράταση μόνο κατά ένα εξάμεινα και μετά θα υπάρξουν νέοι κανόνες βάσει ε, των ε, νέων κανονισμών για τις κρατικές βοήθειες. Δηλαδή θα υποβάλει νέα που τροποποίηση της απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα ισχύουν αυτά σε συνδυασμό με τους κανόνες για τις κρατικές βοήθειες. και έτσι να μπορέσουν και τα κράτη-μέλη να στηρίξουν την ανάπτυξη των ε, μειονεκτουσών περιοχών. Μόνο έξι μήνες λοιπόν για αυτό το λόγο. Η ερώτησή μου είναι, θέλει κάποιος το λόγο, κυρία Μπέντερ. Ευχαριστώ πολύ. Την τελευταία φορά που το συζητήσαμε αυτό με μια έκθεση σχετική, είχα εκφράσει τη δυσαρέσκειά μου σχετικά. Χαίρομαι που μαθαίνω ότι πρόκειται μόνο για μια εξαμηνιαία παράταση. Ε, εσείς τι έχετε καταλάβει, μέχρι να ξαναλλάξουν οι κανόνες θα τα δούμε και εμείς, θα γνωμοδοτήσουμε απλώς ή πάλι απλώς θα ψηφίσουμε. Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση δύο απαντήσεις. Πρώτον, να είναι σαφές ότι πρόκειται μόνο για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τοπικώς παραγόμενα και τοπικώς καταναλωμένα ε, προϊόντα. Ποτά. Δεν μιλούμε για εξαγωγές, αυτό είναι ένα στοιχείο και το δεύτερο είναι ότι η παράταση μόνον έως τον Ιούλιο, Ιούλιο έτσι, ναι, 1η ε, Ιουλίου φέτος ε, σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα απόφαση του Συμβουλίου θα πρέπει να υποβληθεί, ε, αφού προετοιμαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να υποβληθεί και σε εμά, προκειμένου να αποφανθούμε. Οπότε η νέα Επιτροπή Περιφερειών και Περιφερειακής Πολιτικής θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σχέση με τη νέα πρόταση εφόσον ετοιμάζεται τέτοια πρόταση, γιατί θα πρέπει να συνάδει με τους νέους κανόνες που θα έχει εντωμεταξύ θέση σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κρατικές βοήθειες. Ο κύριος Ιράσαμπαλ Μπέιτια. Λίγο βασκικό μου ακούγεται αυτό. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι. Συμφωνήσαμε, συμφωνούμε σε αυτή τη γρήγορη διαδικασία, τη ταχεία και την απλή. Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα. Υποστηρίζουμε την επιτάξη αυτή. Ευχαριστώ. Άρα δεν διαφωνεί κανείς έτσι να το εκλάβω με την απλούστευμένη διαδικασία. Οπότε μπορεί να εγκριθεί αυτό το σημείο με την απλουστευμένη διαδικασία και θετική ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης βάσει του άρθρου 46. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στις ψηφοφορίες σημείων υπαριθμών 7. Να ελέγξουμε τις μηχανές, τα μηχανήματα, ο συνήθως παρακαλώ με τις κάρτες για να ψηφίσουμε, να δούμε αν λειτουργούν. Παρακαλώ ανοίξτε την ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εντάξει, δουλεύουν όλα τα μηχανήματα, πάμε λοιπόν. Ψηφίζουμε. Ε, Η πρώτη έκθεση είναι του Γιουνούς Ομαρζή. Η τροπολογία 29, ο εισηγητής έχει κάνει εδώ μια προφορική, διαφωνεί κανείς με την προφορική τροπολογία, να την ψηφίσουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Νομίζω. Η 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 και 36 μαζί υπέρ. Να ταυτόσιμες κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 40... έλεγχο θέλετε πάμε στη 44 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 29 ειπέ. 7 κατά. 45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 50 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 51 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 52. Τι θέλει αυτό, απάλληψη διαγραφή υπέρ. Ας την ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά τη 52. Πέρας. 17-18 απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 53. Καταπίπτει, αλλά δεν εγκρίθηκε 52, αλλά ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχή. Και πάλι έλεγχο χρειάζεται για την 53. Νομίζω ότι είχε απορριφθεί, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Πέρας. Ναι, όντως απερίφθη. Λοιπόν, πάμε στην 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 56 κατά πίπτη, εφόσον εγκρίθηκε η προηγούμενη συμβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 63 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 64 το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο έλεγχος. Το δεύτερο τμήμα της 64 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απεριφθεί. Η 65 είπε. κατα Κατά αποχές εγκρίνεται. 66-67 μαζί είπε. Κατά αποχές εγκρίνονται. 68 και 69 είπε. Κατά αποχές εγκρίνονται. 70 είπε. Κατά αποχές εγκρίνονται. 71 είπε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 Πέρας. Απορρίπτεται. 78 είπε. Να την ελέγξουμε και αυτή παρακαλώ. 78 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται έτσι σε ισοψηφία έχουμε απόρριψη. 79 είπε. Πάλι έλεγχος για την 79 παρακαλώ. τι έγινε, αλλάξατε γνώμη, συντονιστές, δείχνετε άλλη. Ε, ε, εγκρίθηκε 80 ε, είπε, κατά αποχές εγκρίνεται, 81 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται, 82 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 10 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται, 86 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται, 87 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 11 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται, 80... Όχι, ε, πού είμαστε τώρα, 11 την ψηφίσαμε. Και μετά που πάμε στην 91 τροπολογία, 91 ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 100 υπέρ έλεγχος για την 100 τροπολογία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ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 Ε, μου είπε ο Λάμπερτ Βανίστερο να την υπερψηφίσω, οπότε την υποστηρίζω, τι να κάνω. 135 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται, 136 και 37 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, 138 υπέρ έλεγχος για την 138 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 προς 18. 139 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 145 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 146 και 7 ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 100 πώς απορρίφθηκε. 152 τώρα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 και 5 υπέρ να ελέγξουμε για αυτές τις δύο 154 και 155. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίβεται Ποιε ήταν αυτέ. Α, 156, μάλλον 150. Όχι 157 α, ωραία. 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 να ελέγξουμε για τον 157 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 158. 158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 23 υπέρ. Συμβαστική 3. Με συγχωρείτε, προσπάθησα να κλέψω και δεν τα κατάφερα. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23. Σωστά, υπέρ. Ελέγχουμε για τον 23. Άρχεται η προσφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 24. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ να ελέγξουμε και για τον 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 και 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Τι, Ναι, 31 προς 2. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Ε, Περνάμε τώρα στη γνωμοδότηση του κυρίου Σταυρακάκη. Γνωμοδότηση για την απαλλαγή 2012. Ψηφίζουμε τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η γνωμοδότηση όπως ε, τροποποιήθηκε άρτη ψηφοφορία. 33 υπέρ, επομένως εγκρίνεται. Και ουδής κατά, είχαμε μερικές μόνο αποχές. I don't know whether we already have the... Δεν ξέρω αν έχουμε ήδη στην αίθουσα τους εμπειρογνώμονες για την δημόσια ακρόαση που θα ακολουθήσει. see uh, anybody. Αγαπητοί συναδέλφοι, έχουμε δύο σημαντικά σημεία ακόμα στην ημερήσια διάταξη για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Το πρώτο σημείο έχει να κάνει με την ισότητα των φύλων στις περιφερειακές αυτές πολιτικές και στη συνέχεια έχουμε ένα σημείο για την στρατηγική Αδριατικής Ιωνίου. Περιμένουμε τους εμπειρογνώμονες που θα πάρουν το λόγο. Όταν μπουν στην αίθουσα, ενημερώστε μας να ξεκινήσουμε. You want to speak? Yes, uh, Jan Ο κύριος Ολμπρίχτ, έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας, δεν έχουμε διακόψει. Jan Ολμπρίχτ, ένα ερώτημα. Στο πρώτο τμήμα της συνεδρίασης σας εξήγησα ότι ως μέλος Επιτροπής Προπολογισμών έχω λάβει όλες τις πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, όλες αυτές τις λεπτομερείς πληροφορίες. Νομίζω ότι και εμείς ως μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες. Λέγονται εδώ πέρα τα πάντα όσον αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων, τις πληρωμές κτλ. Ναι, ουσιαστικά πρέπει να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να στέλνουν και σε εμά αυτέ τι πληροφορίε, όχι μόνο στην Επιτροπή Προπολογισμών. Ναι, συμφωνεί ο κ. Όλμπρεκτ. Ναι, λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε το αίτημα αυτό, δηλαδή ό,τι αποστέλλεται στην Επιτροπή Προπολογισμών να αποστέλλεται και στη δική μας την Επιτροπή. Έχεις κάποια ηλεκτρονική εκδοχή αυτών των δεδομένων ώστε να τα λάβουμε. Νομίζω ότι το έχουμε και ηλεκτρονικά το έγγραφο αυτό. Μπορώ να σου διαβιβάσω λοιπόν. Μπορεί να ασχοληθεί με αυτό η γραμματεία και όλα τα μέλη της Επιτροπής μας μπορούν να λάβουν τα στοιχεία αυτά ηλεκτρονικώς και εγώ βέβαια θα μπορέσω να τα λάβω. Where? I will tell that they uh,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 Σας παρακαλώ, σας περιμένουμε. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε συναδέλφους και καλεσμένους που θα παρουσιάσουν την πρωτοβουλία για την δημιουργία μιας νέας Εμβληματική μάλλον πρωτοβουλία για την ισότητα των φύλων στις περιφερειακές πολιτικές για την ανάπτυξη στην περιοχή της Βαλτικής. Έχουμε την Μάρτα Χόζερ Κόσμιελ, την ε, εκπρόσωπο από το Winnet Center of Excellence, κέντρο αριστείας Winnet από το Πανεπιστήμιο του Στέτιν της Πολωνίας. Έχουμε επίσης την Εύα Ρουμίνης Καζίμη από το Διεθνές Φόρουμ Γυναικών Οικονομικής Σχολή της Βαρσοβίας και την Μπρίτ Μαρή Σόντερμπερκ ε, Τόστερστον, πρόεδρος της Ένωσης Γουίνετ Σουηδία. Πρέπει να ξεκινήσουμε, αν δεν κάνω λάθο, η Μπρίτ Μαρή θα πάρει πρώτα το λόγο, παρακαλώ. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνετε να συμμετάσχουμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής σας για να συζητήσουμε και να παρουσιάσουμε ουσιαστικά το ζήτημα αυτό που άπτεται της ισότητας των φύλων στις ε, περιφερειακές πολιτικές για την ανάπτυξη. Η δημιουργία ενός εμβληματικού σχεδίου για την ισότητα των φύλων στην περιοχή της Βαλτικής είναι μια ιδέα που ξεκίνησε με το σχέδιο capitalization του Interreg το 2010 και το 2011 και συμμετείχαν 8 χώρες σε 9 προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας στα βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά της Ευρώπης και επικεντρωθήκαμε στο πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες συστάσεις χάραξης πολιτικής ε, για την ε, Στρατηγική Ευρώπη 2020, για το Περιφερειακό Ταμείο και το Κοινωνικό Ταμείο. Γίνανε οι συστάσεις αυτές που τις βλέπετε στο έγγραφο αυτό με τον πράσινο τίτλο και έχουμε και κάποια θετικά παραδείγματα από όλες αυτές τις περιοχές της Ευρώπης που συμμετείχαν στα προγράμματα αυτά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όλες αυτές οι περιφέρειες υπέβαλαν επίσης και σχέδια δράσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότητα των φύλων στις μελλοντικές περιφερειακές πολιτικές της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οργανισμοί εκπροσώπησης των συμφερόντων των γυναικών, πολιτικοί αλλά και ιδιωτικέ εταιρείε συμμετείχαν στο εγχείρημα αυτό. Η ε, πλατφόρμα εταιρική σχέση της ε, Βαλτικής για την ισότητα των φύλων και την οικονομική ανάπτυξη βασίζεται στα συμπεράσματα αυτά του WINET 8 και θέλαμε να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε στη συγκεκριμένη αυτή περιφέρεια τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα. Και ουσιαστικά επικεντρωθήκαμε στην καινοτομία και την ισότητα των φύλων για την οικονομική ανάπτυξη. Χρησιμοποιήθηκαν κονδύλια από το ειδικών Ινστιτούτο που εκπροσωπώ και συνεργαστήκαμε και με το Διεθνές Φόρουμ Γυναικών καθώς επίσης και με την Σχολή Οικονομικών της ε, Βαρσοβίας, καθώς επίσης και με το Πανεπιστήμιο του Στέτιν της Πολωνίας. Θελήσαμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε τα συμπεράσματά μας στην περιφέρεια της Βαλτικής και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα εταιρικής σχέσης για την ισότητα των φύλων και την οικονομική ανάπτυξη με βάση τα πορίσματα του κέντρου αριστείας Winnet. Ε, Θέλαμε επίσης να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κέντρο πόρων για τις γυναίκες και θα, πώς θα μπορούσε αυτό να συμβάλλει σε ζητήματα όπως η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, οι τεχνολογίες πληροφορικής. Και έτσι, φέτος, καταλήξαμε στην ιδέα της δημιουργίας μιας ε, εμβληματικής πρωτοβουλίας ενός flagship project συγκεκριμένα για την περιφέρεια αυτή και αυτό που φασίστηκε μάλιστα το 2013 στην Βαρσοβία. Η Λιθουανία, η Εστονία και η Λετωνία συμμετέχουν, καθώς επίσης και η Γερμανία και η Δανία. Ο γενικότερος στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση της ευημερίας, ένας επιμέρους στόχος είναι να καταφέρουμε να συμβάλλουμε στην περαιτέρω πρόθεση της ε, ε, στρατηγικής για την περιφέρεια της ε, Βαλτικής και πώς μπορούμε να πετύχουμε περισσότερο τους στόχους της Ευρώπης 2020. Και όσον αφορά τους γενικούς τρομείς προτεραιότητας, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η κοινοτομία και η εμπλοκή όσο δυνατόν περισσότερων παραγόντων. Ένα επιμέρου στόχο θα πρέπει να είναι να προωθηθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, καθώ επίση και τα προγράμματα τα εκπαιδευτικά, καθώ επίση και κάποιοι γενικότεροι στόχοι όσον αφορά την τεχνολογία τη πληροφορία και των επικοινωνιών. Θέλουμε να καταφέρουμε να επανακαθορίσουμε κάποιες πολιτικές όσον αφορά την καινοτομία και να συνδυάσουμε πλέον κοινωνική και τεχνολογική διάσταση από τη σκοπιά της ισότητας των φύλων. Θεωρούμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε καλύτερους πλέον ορισμούς και καλύτερες προτάσεις. Θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει να υποβληθούν κάποιες συστάσεις καθώς επίσης και ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε περισσότερο τη διάσταση του φύλου στην βιώσιμη σε μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα προωθεί την κοινοτομία πάντα για την περιφέρεια αυτή της Βαλτικής. Θέλουμε επίσης να επικεντρωθούμε όσο δυνατόν σε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάνουμε λοιπόν κάποιες συστάσεις για την χάραξη πολιτικής προκειμένου να καταφέρουμε να ε, συνδυάσουμε περισσότερο, να ενσωματώσουμε μάλλον περισσότερο την ισότητα των φύλων σε όλες τις σχετικές στρατηγικές και δράσεις για την περιφέρεια της Βαλτική. Θεωρούμε ότι το σχέδιό μας αυτό θα μπορέσει να αποτελέσει πρότυπο, αφού δοκιμαστεί στη δική μα την περιφέρεια, θα μπορέσει να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες μακροπεριφέρειες και σχετικές στρατηγικές. Με άλλα λόγια, θέλουμε αυτή η εμβληματική πρωτοβουλία, αυτό το flagship project, να αρχίσει να εφαρμόζεται και σε άλλες περιφέρειες. Η πρώτη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στην Στοκχόλμη, στη Σουηδία, στις 27 Φεβρουαρίου του 2014 και θα επικεντρωθούμε στα ζητήματα τη οικονομική ανάπτυξη και τη ισότητα των φύλων πάντα στα πλαίσια αυτή τη πλατφόρμα εταιρική σχέση για τη Βαλτική. Στη στρατηγική τη Βαλτική ήδη λέγεται ότι η σε εφαρμογή της στρατηγικής απαιτεί επίσης την έγκριση της διάστασης της ισότητας των φύλων στο σύστημα διακυβέρνησης και στο σχέδιο δράσης. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί κεντρικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, μπορούν να προκύψουν οικονομικά ωφέλη και ωφέλη για τις επιχειρήσεις εφόσον καταφέρουμε να ενισχύσουμε τη διάσταση της ισότητας των φύλων. Προκειμένου να πετύχουμε τους βασικούς στόχους της μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη Βαλτική θα πρέπει να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε και τη συμβολή αλλά και τα πολλά προσόντα και ταλέντα τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών. Αυτό λέγεται επισήμως αυτή τη στιγμή στο κείμενο της στρατηγικής μας. Ευχαριστώ. Good afternoon. Καλησπέρα σας. Το όνομά μου είναι Μάρτα Χόζερ Κότσμιλ και εκπροσωπώ το Πανεπιστήμιο του Θετσίν από την, το τμήμα της οικονομίας και της, του management και στατιστικής. Από το, 2010, από το 2004 συνεργαζόμαστε με το Βίνετ της Σουηδίας και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο δημιουργίας του κέντρου αριστείας του Βίνετ για τις χώρες της Βαλτικής. Μετά από πέντε ημέρες ε, συνομιλιών για τη σχέση ισότητας και ανάπτυξης δεν θα είχαμε καταλήξει σε συμπέρασμα. Όμως θα ήθελα να σας ε, πω κάποιες από τις δικές μας βασικές ιδέες. Στόχος της παρουσίασής μου θα είναι να σας δείξω τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης και της ισότητας των φύλων στην περιοχή των χωρών της Βαλτικής. Από το 1995 έως το 2012 παρατηρούμε μια σαφή σταθερή αύξηση του ΑΕΠ ανακεφαλής στην εικόνα στα αριστερά ενώ στην εικόνα στα δεξιά βλέπουμε τα ποσοστά ανάπτυξης του ΑΕΠ. Βλέπουμε μεγάλη πτώση ε, λόγω της διεθνούς κρίσης. Στην πλειονότητα των χωρών της Βαλτικής, ο δείκτης της ισότητας των ε, φύλων ε, γνώριζε σταθερή αύξηση παράλληλη. δηλαδή υπήρχε καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος της ισότητας των φύλων. Και αυτό το σημείωσε και η UNDP. Είδαμε μάλιστα κάποια μείωση το 2010 σε σχέση με το 2005 σε ορισμένες χώρες. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η Πολωνία και η Λετωνία λόγω του χαμηλότερου ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ως αποτελέσμα της κρίσης. Εάν συγκρίνουμε αυτές τις δύο διαστάσεις, δηλαδή την ανάπτυξη και την ισότητα των φύλων και τους δείκτες τους, θα παρατηρήσουμε μια ισχυρή και θετική ε, εξίσωση, έναν αλληλοσχετισμό μεταξύ της ισότητας των φύλων και της αύξησης του ΑΕΠ ανακεφαλή. Με συγχωρείτε, είναι σαφής αρνητική η εξίσωση. Δηλαδή, όσο πιο πολύ αυξάνεται η οικονομία, τόσο χαμηλότερα είναι τα ποσοστά ε, του άλλου δίκτυ. Ενώ είναι θετική η εξίσωση, ο συσχετισμός δηλαδή, της ισότητας των φύλων σε συνάρτηση με το ανακεφαλή ΑΕΠ. Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις χώρες της Βαλτικής σε δύο ομάδες. Πρώτα απ' όλα ως προς το υψηλό εισόδημα και το χαμηλότερο. Εκεί δηλαδή που οι γυναίκες συμβάλλουν πολύ λιγότερο στην ανάπτυξη από ότι οι άντρε. Γιατί συμβαίνει αυτό σε αυτές τις χώρες χαμηλών εισοδημάτων. Μια από τις απαντήσεις είναι λόγω των διαφορών στην κατανομή του χρόνου. Δηλαδή, στη διαφάνεια βλέπετε τη χρήση χρόνου ανά τον προϋπολογισμό στις περιοχές στην περιοχή των χωρών της Βαλτικής. Βλέπουμε ότι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι γυναίκες περνούν περισσότερο, λιγότερο χρόνο στην αμοιβόμενη εργασία από ότι άνδρες και πολύ περισσότερο στην μη αμοιβόμενη. Δηλαδή έχουν λιγότερο ελεύθερο χρόνο από ότι άνδρες. Άρα προτείνουμε το εξής ένα κανόνα με τρία ρο στα αγγλικά, δηλαδή να, επανα, να επανεξετάσουμε την έννοια της αμοιβόμενη και μη αμοιβόμενη εργασίας, να καταγράψουμε τον όγκο της αμοιβόμενη και μη αμοιβόμενη εργασίας και να ξανακατανείμουμε την ε, μη αμοιβόμενη εργασία μετατρέποντάς τη σε αμοιβόμενη στην αγορά εργασίας. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια από τις αποκρίσεις μας για την αντιμετώπιση της κρίσης και για να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη στην περιοχή των χωρών της Βαλτικής. Αυτό ήταν μόνο ένα παράδειγμα από μια από τις έρευνες που έγιναν από το WinNet ω κέντρο αριστείας είναι πολύ καλό που μπορούμε να δουλέψουμε για έναν τόσο ε, αποτελεσματικό οργανισμό όπως το WINET της Σουηδίας αλλά μπορούμε να συνεργαστούμε και με άλλους ε, σοβαρούς εμπειρογνώμονες όπως η Εύα Τζίμνη και να πω δύο λόγια για το κέντρο μας. Το κέντρο αριστείας του Winnet είναι ένα κέντρο από το Διεθνές Δίκτυο Ερευνητών για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας με σκοπό να καταρτήσει και να προωθήσει την έρευνα, τη διδασκαλία και την χάραξη πολιτικής για την ισότητα των φύλων, την κοινοτομία και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που έχω να σας μιλώ. Λέγομαι Εύα Ρουμίνσκα Καζίμνη από το Διεθνές Φόρουμ Γυναικών που είναι γυναίκες πανεπιστημιακές και επιχειρηματίες, κυρίως ε, δραστηριοποιούνται στον χώρο της οικονομίας. Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος περιφερειακής πολιτικής στην ανάπτυξη, στις θέσεις εργασίας και στην οικονομία, χρειάζονται τουλάχιστον δύο πράγματα. Να χρησιμοποιηθεί αυτή η ιδέα της μακροπεριφέρειας, που είναι μια καινούρια έννοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεύτερον, να ενταχθεί και η διάσταση του φύλου που λείπει από τις στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης και περιφερειακής πολιτικής δούμε λοιπόν και επιλέξουμε να ακολουθήσουμε τις μακροπεριφέρειες, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η πρώτη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ε, Βαλτική θάλασσα κατανοεί ότι η μακροπεριφέρεια είναι κάτι που συμβαίνει στη ζωή συνεργάζονται περιφέρειες μεταξύ τους και στην Ανατολική Ευρώπη και στο Δούναβι χωρίς να υπάρχει καμιά τεράστια στρατηγική. Από μόνη της η ζωή το φέρνει. Ε, αν δείτε ε, τους βασικούς στόχους ε, αυτής της στρατηγικής είναι η ανάπτυξη και η καινοτομία. Και εγώ προσπαθώ να πω ότι δεν έχει ενταχθεί η διάσταση του φύλου είναι ακόμα μια διαδικασία εκμάθησης, βλέποντας και κάνοντας δηλαδή, αλλά ε, παραμένω εγώ στην ιδέα μου ότι το μοντέλο ε, έχει πλέον ανοίξει την πόρτα για μια νέα προσέγγιση και δίνει και το καλό παράδειγμα για εθνικές στρατηγικές και τις τοπικές και τις περιφερειακές ως προς τη διάσταση του φύλου. Λέμε λοιπόν ότι μόλις άνοιξε η πόρτα, μια χαραμάδα είναι, δεν είναι καμιά ανοιχτή θύρα. Υπάρχει ε, ένα στοιχείο που ανέφερε η προλαλήσασα, αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι τομέας προτεραιότητας και υπάρχει αυτή η διάσταση για το στοιχείο του φύλου. Σε πολλούς άλλους τομείς όμως αυτή απουσιάζει και αυτό γιατί δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις και επιχειρησιακά προγράμματα που να εντάσσονται στη στρατηγική αυτή. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα, είναι επίκαιρο το θέμα να ενταχθεί στο σχέδιο. Αυτό συζητούμε άλλωστε. Αν δείτε ε, τον παράγοντα γυναίκα στην ανάπτυξη, ε, το αναγνωρίζουν πολύ πλέον, είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι γυναίκες είναι νέα πηγή εργασίας, είναι και το οικονομικό επιχείρημα αλλά και το επιχείρημα της διαφοροποίησης ε, για την καινοτομία και την προληπτική προσέγγιση. Δεν μπορεί κανείς να έχει μια ευφυή ή καινοτόμα οικονομία, ευφυή τη λέμε τώρα, που να κυριαρχείται από την ε, προσέγγιση των ανδρών. Χρειάζεται διαφοροποίηση. Και τέλος το επιχείρημα που είναι αρκετά σαφές είναι ότι η Ευρώπη όπως είπε και η Επίτροπος Βίβιαν Ρέντι, δεν μπορεί να ε, αν έχετε πλέον την κατάσταση που να έχει τις πιο μορφωμένες νοικοκυρές. Οι γυναίκες είναι πάρα πολύ μορφωμένες με πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο και πάει χαμένη αυτή η γνώση όταν ασχολούνται με τα οικιακά η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 θα πρέπει να ε, αναβαθμίσει τις υποβαθμισμένες περιφέρειες. Εκεί θα καταλάβουμε ότι η γεννητήρια δύναμη είναι οι γυναίκες. Στη Σιλεσία της Πολωνίας που είναι μια περιοχή με ανθρακοριχία, και εκεί κυριαρχεί ε, ο γυναικείος πληθυσμός, είναι πάνω από το 45% γιατί οι άνδρες έχουν φύγει ε, για να βρουν δουλειά αλλού. Και κυριαρχούν και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι γυναίκες, στον τουρισμό γενικότερα. Αν δούμε τις στρατηγικές τώρα, είτε αυτές είναι μεγάλες, στρατηγική δια του 2020 ή απλώς τοπικές για την περίοδο 2014-2020, θα διαπιστώσουμε ότι πολύ λίγα στοιχεία έχουν σχέση με το φύλλο. Και εμείς στο Κογκρέσο των ε, ε, Λονών Γυναικών έχουμε εκπονήσει μία μελέτη, αναλύσαμε την κατάσταση και διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει διάσταση φύλου. Και όταν ε, κοιτάς μια περιφέρεια και τις αδυναμίες της, χρειάζεται αυτή η έξυπνη εξειδίκευση αλλά χρειάζεται να βάνονται υπόψη και αυτά τα στοιχεία του φίλου. Αν με ρωτήσετε τώρα γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη, ο κρίκος που λείπει από τη στρατηγική, βασικός λόγος είναι ότι η ισότητα του φίλου θεωρείται κάτι άσχετο με την οικονομία. Θεωρούν οι οικονομολόγοι ότι είναι ουδέτερη προς το φύλλο η οικονομία. Όταν εκπονούν αυτές τις στρατηγικές δεν το θεωρούν ως ένα τμήμα φυσικό της στρατηγικής. Ότι η οικονομία είναι ουδέτερη, δεν έχει φύλλο. Αν δείτε λοιπόν τις στρατηγικές έχουν κάποια στοιχεία, κάποιες συνιστώσεις φύλλου που έρχονται να προσθεθούν με τρόπο πάρα πολύ τεχνητό σε όλη τη στρατηγική σε διάφορα επίπεδα. Αυτό δεν ενσωματώνει τα θέματα από την αρχή και την ε, διάσταση του φίλου, Όχι μόνο στην αφήγηση γενικά της στρατηγικής, αλλά και στο ε, επιχειρησιακά προγράμματα, στους δείκτες επιτυχίας. Για παράδειγμα, στην Πολωνία εμείς έχουμε ένα δείκτη για τη δημιουργία ε, θέσεων εργασίας σε μια επαρχία. Αλλά εκεί δεν αναφέρεται η κατανομή ένα φύλλο. Πόσες θέσεις δημιουργήθηκαν για γυναίκες, πόσες για άντρες, πώς ε, προωθείται το επιχειρηματικό πνεύμα. Είναι απλώς ε, συνολικά νούμερα. Δεν υπάρχει αυτή η κατανομή. Και αυτό έχει συνέπειες όμως για το πώς θα κατανέμονται οι πόροι και πώς θα χρηματοδοτούνται τα προγράμματα. Και έχουμε δει ότι αυτό δεν δούλεψε πάρα πολύ καλά την προηγούμενη ε, προγραμματική περίοδο που 7 με 8% των έργων των project είχαν πραγματικά ένα στοιχείο φύλου με στρατηγική και με χρηματοδότηση συνδυασμένη. Άρα είναι σημαντική διάσταση του φύλου, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στις στρατηγικές που εκπονούμε, στην οικονομία. Και επίση μιλούν πολύ διαφορετική γλώσσα οικονομολόγοι και εκείνοι που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων. Είναι λίγο παράλληλες αυτές οι συζητήσεις. Ε, δεν χρησιμοποιούν ούτε την ίδια γλώσσα, ούτε τι ίδιε έννοιε. δεν έχουν κοινή πλατφόρμα για να συνεννοηθούν. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία του κάθε έργου για τη Βαλτική θάλασσα είναι να δημιουργηθεί μια τέτοια πλατφόρμα σε μεγάλο επίπεδο αυτό της μακροπεριφέρειας για να μπορούν οι διάφορες ομάδες να συζητούν και να καταλήγουμε μια συναντήληψη και μια κοινή γλώσσα. Και βέβαια είναι λίγε οι γυναίκε σε, επίπεδα λήψη αποφάσεων. Καλό θα ήταν να αυξηθεί ο αριθμό του. Είναι προφανέ, δεν χρειάζεται να επεκταθώ σε αυτό. Μόνο 3% είναι πρόεδροι σε δυτικά συμβούλια εταιριών οι γυναίκες. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Τελειώνω με τις προκλήσεις για το περίοδο 2014-2020. Βασικό είναι να υπάρχει έρευνα στραμμένη προς ε, τη συγκεκριμένη πολιτική και στις διαστάσεις του φύλου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα το καταλάβουμε, πώς θα συνδέσουμε την ισότητα με την καινοτομία και την ευφυή οικονομία στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας. Ε, στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργηθούν αυτές οι εταιρικές σχέσεις και να αρχίσει ένας διάλογος μεταξύ διαφόρων ε, φορέων, πρωταγωνιστών και να ε, δούμε ποιοι είναι οι δείκτες επιτυχίας μιας στρατηγικής με βάση το φύλλο και να βοηθηθούν οι χώρες να κάνουν ειδικές συστάσεις και δράσεις. Και νομίζω ότι το πρόγραμμα, το έργο που σας παρουσιάζουμε τώρα και το κέντρο αριστείας Γουίνετ θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Μετά από αυτή την τριετία που είναι το προπαρασκευαστικό στάδιο, ελπίζουμε να έχουμε καταλήξει σε απορίσματα για να τα μοιραστούμε με άλλες περιφέρειες, όπως είναι η Νότιο-Ανατολική Ευρώπη ή η περιφέρεια του Δουνάβιου. ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Όλμπρεχτ έχει το λόγο πρώτος. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Θα σας μιλήσω λοιπόν στα πολωνικά. Καθότι προέρχεστε από τη χώρα μου. Μία ερώτηση και δύο παρατηρήσεις. Μπορείτε καταρχάς να διευκρινίσετε ένα σημείο Πώς κατανοείτε εσείς το ζήτημα της αμοιβόμενη και μη αμοιβόμενη εργασίας. Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένες για το σημείο αυτό. Επίσης, πώς συσχετίζονται αυτές οι δύο έννοιες αμοιβόμενη και μη αμοιβόμενη εργασία στην παρουσία στην οποία κάνατε. Πρώτον αυτόν. Δεύτερο, ένα ερώτημα το οποίο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση τέλος πάντων με το ερώτημά μου αυτό. Αναφερθήκατε περισσότερο στις γυναίκες, προσεγγίσετε τα πράγματα από τη σκοπιά των γυναικών. Τι γίνεται όμως με τους άντρες. Αναφερθήκατε σε κάποια επαγγέλματα τα οποία είπατε ότι είναι κυρίως γυναικεία. Το θέμα είναι να μπορούν και οι άντρες να έχουν πρόσβαση όμως στα επαγγέλματα αυτά δεν παρεμποδίζεται η πρόσβασή τους. Δεν λέω αυτό το πράγμα, αλλά μήπως θα πρέπει να εξελιχθεί κατά κάποιο τρόπο η ίδια η φύση των επαγγελμάτων αυτών, ώστε να απευθύνονται πιο εύκολα και στους άνδρες και στις γυναίκες. Ξέρετε ότι ένα άλλο ζήτημα τώρα, μιλάμε για μακροπεριφερειακές στρατηγικές, όχι μόνο στην, περι... στην περιφέρεια της Βαλτικής. Πιστεύω ότι γενικότερα στην ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ισότητα των φύλων και ορισμένες φορές αντιμετωπίζουμε κάποια αυθαίρετα τεχνητά προβλήματα. Για παράδειγμα, στα ερωτηματολόγια που έχουμε για τα επιμέρους έργα υπάρχει ένα ερώτημα, το ακόλουθο. Αιτιολόγηση διαφόρων στοιχείων που καταδεικνύουν ότι όντως υφίσταται ισότητα των φύλων στα προγράμματα αυτά, στα έργα αυτά. Πολλές φορές οι απαντήσεις που μας δίνονται είναι πολύ επιφανειακές. Παρ' όλα αυτά οι απαντήσεις όμως είναι σημαντικές γιατί μπορούν να επηρεάσουν το ίδιο το έργο και την εικόνα του έργου, την προβολή του έργου αυτού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι επιφανειακές αυτές απαντήσεις μπορεί να αποβούν ιδιαίτερα επιζήμιες. Στην Σιλεσία, στην οποία αναφερθήκατε, Όντως ακολουθείται ένα ιδιαίτερα πατριαρχικό μοντέλο. Οι περισσότερες γυναίκες όντως μένουν στο σπίτι και ασχολούνται με τα οικιακά και έχει προκύψει μια πραγματική ανάγκη εμπλοκή των γυναικών στην αγορά εργασίας για να αντιμετωπιστούν διάφορες προκλήσεις πλέον και προβλήματα που έχει αυτή η περιοχή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν κατασκευάζουμε ένα αυτοκινητόδρομο, Ξέρετε ότι θα πρέπει να εργαστούν για το έργο αυτό τόσο άντρες όσο και γυναίκες. Και βέβαια τον αυτοκινητόδρομο αυτό συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν και άντρες και γυναίκες. Πολλές φορές όταν έλεγα για αυθαίρετες απαντήσεις, μας λένε όταν απαντούν στο ερωτηματολόγιο ότι κοιτάξτε, όντω τηρείται η ισότητα των φύλων για το συγκεκριμένο αυτό έργο, ακριβώ επειδή και άντρε και γυναίκε θα χρησιμοποιήσουν το έργο αυτό εν προκειμένου τον αυτοκινητόδρομο. Ξέρετε ότι αυτό δεν αρκεί. Ο κύριος Νίλσον έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εγώ τη μητρική μου γλώσσα. Ένα ερώτημα καταρχάς θέλω να θέσω. Όταν μιλάμε για τέτοια εμβληματικά έργα σε μακροπεριφερειακό επίπεδο, νομίζω ότι ένας στόχος θα πρέπει να είναι πάντα να χρησιμοποιούμε την εμπειρία την οποία έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε περιφερειακό πλέον επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να εμπλουτίσουμε τα έργα αυτά με την εμπειρία που έχουμε ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βάσει της δικής μου τώρα εμπειρία στη Βόρεια Σουηδία, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι όντως αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στη δεκαετία του 90, στη δική μου την περιφέρεια, για έξι περίπου χρόνια, εφαρμόσαμε ένα σχέδιο το οποίο είχε ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερο την γυναική επιχειρηματικότητα και τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ θετικά και είδαμε στη συνέχεια ότι τα αποτελέσματα του έργου αυτού Στη συνέχεια τροφοδότησαν, εμπλούτησαν και άλλα έργα τα οποία εφαρμόστηκαν στη δική μου την ε, περιφέρεια. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες οι οποίες στείνουν κάποιες μικρές επιχειρήσεις τελικά δημιουργούν επιχειρήσεις πιο βιώσιμες από αυτές που δημιουργούν οι άντρες. Και επίσης βλέπουμε ότι οι γυναίκες μεταξύ τους ε, δείχνουν μεγαλύτερη ελεγγύη από ότι οι άντρες οι γυναίκες επιχειρηματίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές θετικές επιπτώσεις και εν τέλει το αποτέλεσμα γενικεύεται έπειτα. Και κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και η οικονομική ανάπτυξη σε όλη την περιοχή. Ευχαριστώ κύριος Βανίστερο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίο είναι που συζητούμε αυτό το θέμα της Βαλτικής θάλασσας να ακούμε και τις θέσεις και την προσέγγιση κυρίως ε, ε, των γυναικών και να κοιτάμε και τα θέματα φύλου. Έχω μια ερώτηση εγώ που έχει να κάνει με την προσέγγιση στα διάφορα κράτη-μέλη. Είναι μια ευρύτερη περιφέρεια, οι βαλτικοί χώρες εντός ένωσης, εκτός ένωσης. Στη στρατηγική αυτή συμμετέχουν οι χώρες και δεσμεύονται να κάνουν κάποια βήματα. Θα μπορούσατε εσείς να μας πείτε πώς έχει αυτή η συνεργασία στο δικό σας κέντρο και αν είναι δεσμευτική, δηλαδή αν υποχρεούται κάποιος που συμμετέχει σε αυτή να ακολουθήσει κάποια βήματα. Και εδώ σκέφτομαι και την εκπαίδευση και την κατάρτιση που είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα και δυνατότητες να έχουν περισσότερες ευκαιρίες ε, τα δύο φύλλα. Μπορείτε να εμβαθύνετε λίγο σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σικό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν σας κρύβω ότι βρίσκω ότι εδώ υπάρχει κάποια ασάφεια. Ως Πολωνός είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που έχουμε εδώ Πολωνές ε, εκπροσώπους, ομιλήτριες. Και είναι πολύ ωραίο το όλο εγχείρημα που μας παρουσιάζουν. Από την άλλη όμως βρίσκω ότι το όλο θέμα που μας απασχολεί διέπεται από ασάφεια. Η μεγαλή, το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας στην Πολωνία αναρωτιέται αναρωτιέται για πολλά ζητήματα. Βεβαίω είναι υπέρ τη ε, ένταξη τη Πολωνία και τη συμμετοχή τη Πολωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ψηφίσαν στην Πολωνία εδώ και χρόνια. Όμω δεν είναι αυτό μόνον. Νομίζω ότι οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Ρόμπερτ Σούμαν θα πρέπει να τρίζουν τα κόκαλά τους στους τάφους τους αν βλέπουν τι γίνεται σήμερα. Η ελευθερία της κυκλοφορίας, η ελευθερία των εργαζομένων και των αγαθών, προϊόντων και επενδύσεων. Δεν είναι ιδέες μόνον ιδανικά. Είναι αρχές οι οποίες φαίνεται ότι δεν εφαρμόζονται 100% στην πράξη. Εγώ θέλω να είμαι και ρεαλιστής και να είμαι και ε, υπερασπιστής του ευρωπαϊκού ιδεόδους, αλλά όχι με υπερβολικό ενθουσιασμό. Δηλαδή, τα κριτήρια για την ισότητα των φύλων μέσα από την περιφερειακή πολιτική, την πολιτική συνοχή στις χώρες της περιοχής της Βαλτικής, και το πόσο συμβάλλουν στην πολιτική συνοχή. Δεν νομίζω ότι εμεί έχουμε τον τρόπο να επηρεάσουμε. Νομίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι γυναίκες να έχουν ε, την ε, χαρά να εξελιχθούν μέσα από τη σταδιοδρομία του, να έχουν σωστέ ε, άδειε μητρότητα, οι αμοιβέ του να είναι ικανοποιητικέ. Γιατί όμως μια Πολωνή λόγου χάρη πολίτης στο Ηνωμένο Βασίλειο με δυόμιση κατά μέσο όρο παιδιά και φτάνει τελικά να έχει πιο πολύ αριθμικό οικογένεια από ότι στην Πολωνία με 1,5 κατά μέσο όρο παιδιά. στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πάρει 500 στερλίνες αναπαιδί, ενώ ίσως 25 σλότι αναπαιδί στην Πολωνία. Είναι τεράστια λοιπόν η διαφορά στα επιδόματα. Δεν υπάρχει οικονομική υποστήριξη. Εγώ ε, είμαι μηχανικός από το Πτάνσκ, τον Τάντσιχ, στο νότο, στην νότια πλευρά της Βαλτικής. Πιστεύω ότι στη λεκάνη της Βαλτικής δεν περιμένουν αυτό οι άνθρωποι. Χρειάζονται ίσες ευκαιρίες για να εξελιχθούν. Τώρα τον επιβάλλουμε εμεί κανόνες τελείως θεωρητικούς ή βασισμένους σε ιδεολογίες ε, για την συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία είναι άλλο θέμα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο, όμως να συμπληρώσω κι εγώ κάτι σε σχέση με όσο είπε συνάδελφος. Οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να μας δώσουν ε, ένα οικονομικό δυναμικό που δεν αξιοποιείται ακόμη επαρκώς. Σίγουρα η διαφορά δεν είναι μόνο τα 25 ή 500 ευρώ επιδόματος. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λίγα λόγια για να στηρίξω αυτό που έλεγε Μάρτα Χόζερ, ο Κόσμιλ. Ε, η στρατηγική για τις χώρες της Βαλτικής υποστηρίχθηκε και την ασπάστηκαν όλες οι χώρες της περιοχής της Βαλτικής διότι ουσιαστικά εκφράζει κάποιες οριζόντιες αρχές μεταξύ των οποίων και ισότητα των φύλων. Και κατά αυτή την έννοια υλοποιήθηκε αυτή η στρατηγική στις χώρες της Βαλτικής. Είναι κάτι που το ζήτησε και το υποστήριξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν συντάξαμε το πρόγραμμα δράσης υπήρξαν κάποια πρώτα σχέδια και προγράμματα, ιδίως ένα που το ε, υποστήριξε με εκπαιδευτικού στόχους, Εκεί ήταν ένα από τα πρώτα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί στο πρόγραμμα δράσης, το Quick Equal όπως ονομάστηκε. Υπήρξαν και άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται και θα πρέπει βεβαίως και υπεύθυνη της στρατηγικής για την υλοποίηση, υπεύθυνη για την υλοποίηση της στρατηγικής να αναλάβουν δράση για τόμους όπως η κοινοτομία, η εκπαίδευση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προσπαθούμε εδώ κάπως να ομαδοποιήσουμε τις αρμοδιότητες που θα αναλογούν στον καθένα για να αντιμετωπίσουμε και τέτοιου είδους ζητήματα. Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την ίδια την διοίκηση, το πώς αυτά τα προγράμματα υλοποιούνται στην πράξη. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή συντάσσεται και κατά πάσα πιθανότητα θα δημοσιευτεί μια ανακοίνωση για την ε, για τις στρατηγικές των μακροπεριφερειών, τις οποίες θα πρέπει να τις υλοποιούν και την ευθύνη τους να αναλαμβάνουν οι χώρες τις οποίες, οι οποίες τις ζήτησαν. Το ζήτημα λοιπόν αυτό θα καλύπτεται από την άποψη της μεγαλύτερης ανάληψης ευθύνης για αυτή τη στρατηγική από τους δικαιούχους, από τους παραλήπτες της ε, τρόπον τεινά. Δηλαδή, τα επίπεδα ε, διακυβέρνησης, η ανάληψη ευθύνης είναι κάτι που είναι σημαντικό θα υπάρξει πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέτοιου είδου οριζόντια θέματα να τα αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο στου διάφορου τομεί. Νομίζω το ετήσιο φόρουμ δίνει μια ευκαιρία για συζητήσει, για αφορμέ συνεργασία και για να υποβληθούν προτάσεις για τέτοιου είδου θέματα. Στο τελευταίο ετήσιο φόρουμ στο Βίλνιους παρευρεθήκαμε κι εμείς και όντως είδαμε ότι εκεί σωστά αναφέρουν οι μεν και οι δε τις ανησυχίες τους, προσπαθούν να συμπεριλάβουν στην όλη συζήτηση ε, τα θέματα που πρέπει να επιληθούν. Είναι μια καλή ευκαιρία τέτοιου είδου φόρα και ενθαρρύνουμε όλου να συμμετάσχουν στα δυνατόν περισσότερα στι διάφορε συναντήσει που διοργανώνονται, προκειμένου να εξεταστούν τέτοιου είδου ζητήματα. Ο τρόπος επίσης που μεταδίδουμε τα αποτελέσματα των πιλωτικών προγραμμάτων στη Βαλτική, στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής, είναι σημαντικός. Δηλαδή για να λειτουργήσουν αυτές οι στρατηγικές πρέπει τα διδάγματα που αντλήσαμε από τα διάφορα προγράμματα να ε, γνωστοποιούνται επαρκώς. Και αυτό είναι σημαντικό και για το μέλλον, για να υπάρξει καλύτερο συντονισμός μεταξύ των ε, διαφόρων ε, ε, στρατηγικών μακροπεριφερειών. Υπάρχουν τέσσερις για την ώρα, αυτή της Βαλτικής, της Αδριατικής, του Δούναβη και των Άλπων. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το οριζόντιο θέμα να διέπει όλες τις μακροστατηγικές μας και όχι μόνο να αναφέρεται ε, στα ευρωπαϊκά προγράμματα που προκύπτουν και συσχετίζονται με την πολιτική συνοχή. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Να ζητήσω από του συναδέλφου από το Βίνετ να απαντήσουν. τις κυρίες από το Βίνετ να μας δώσουν τις απαντήσεις τους. Να ξεκινήσω εγώ να σχολιάσω με αυτά που είπε ο Την ερώτησή του. Να απαντήσω ότι το πιο σημαντικό από όσα κάνουμε είναι η ισότητα των φύλων να περάσει και στην πράξη. Δηλαδή να διαδοθεί η εμπειρία μας στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να γίνει κάτι το οικείο σε όλες τις ε, χώρες της περιοχής της Βαλτικής αλλά και στις υπόλοιπες ε, με, με, μακροπεριφέρειες όπως έχουν ονομαστεί στο μέλλον. Βεβαίω έχουμε επαφέ ήδη με του εκπροσώπου και του υπευθύνου τη ε, στρατηγική του Δούναβη για να υπάρξουν οι σχετικέ διαπαθέ. Μάλιστα, οι στρατηγικέ αυτέ έχουν υποστηριχθεί από την Πολωνία και τη Σουηδία σε κρατικό επίπεδο, ώστε να βεβαιωθούμε ότι τη δουλειά μας μπορούμε να την κάνουμε πράξη, να υπάρξει ισότητα των φύλων στην περιοχή της Βαλτικής και γενικότερα τελικά στην Ευρώπη. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Αναφέραμε την εκπαίδευση και τέθηκε μια ερώτηση για το πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι κάθε θεματικός τομέας που συμπεριλαμβάνεται στην στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 και τη στρατηγική για τις χώρες της Βαλτικής, πώς μπορεί να λάβει υπόψη αυτή τη διάσταση καθώς και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, των περιφερειακών αρχών για την εκπαίδευση, δηλαδή από τα δημοτικά σχολεία ως τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πώς στο μέλλον τα μικρά αγόρια και κορίτσια μεγαλώνοντας θα διαλέγουν ελεύθερα τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον, ποια θα είναι η επαγγελματική του ζωή και όχι βάσει των στερεοτύπων των φίλων. Δηλαδή να διαλέγουν αυτό που νομίζουν ότι θα έπρεπε να διαλέγουν αναλόγως με το αν είναι άντρες ή γυναίκες. Αγόρια η νοοτροπία πρέπει να περάσει και στο εκπαιδευτικό σύστημα. E, ja jako statystyk chciałabym się odnieść, e, podzielić kilkoma... Για... Για τα στατιστικά στοιχεία που ζητήσατε, να σας πω και εγώ κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Για την αμοιβόμενη και μια αμοιβόμενη εργασία. Τι σημαίνει ακριβώς. Μιλάμε για την εργασία στην αγορά εργασίας, αυτή είναι η αμοιβόμενη, ενώ η μη αμοιβόμενη είναι η κατοίκον εργασία. Υπάρχει πραγματικά ε, τεράστια απόσταση στον όγκο τη μια και τη άλλη κατηγορία, για τι γυναίκε ιδίω. Όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκε ε, περνούν περισσότερο, πολύ περισσότερο χρόνο στον νοικοκυριό στην ουσία. Ε, Στι δουλειέ του σπιτιού. Στη μία αμοιβόμενη εργασία. Αυτό έχει αντίκτυπο και στο, στα δημοσιονομικά. Όλε οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εκπονούν ένα, ένα σχέδιο προπολογισμού και ακριβώ εκεί βασίζεται και η σύγκριση που κάνουμε για τον κανόνα των τριών ρο ε, στα αγγλικά. Θα πρέπει να ξαναδούμε πραγματικά την έννοια της αμοιβόμενης και αμοιβόμενης εργασίας. Τα επαναλαμβάνω. Έπειτα πρέπει να καταγράψουμε το τι προκύπτει για την αμοιβόμενη ή μια αμοιβόμενη εργασία από τον προπολογισμό και έπειτα να ε, φροντίσουμε και οι άντρες να αναλάβουν ευθύνε στις οικιακές εργασίες για το όφελος και των μεν και των δε. Το αποτέλεσμα της μελέτης μας είναι ότι όσο περισσότερο οι άντρες αναλαμβάνουν κάτι και στο σπίτι, τόσο περισσότερο οι χώρε έχουν ισορροπημένη κοινωνική ζωή. Αυτό το διαπιστώνουμε στι χώρε τη Βαλτική τουλάχιστον. Ε, πρέπει να βρούμε διέξοδο από την κρίση και γι' αυτό ακριβώ πρέπει να ενθαρρυνθούν γυναίκε να δραστηριοποιηθούν στην αγορά εργασία. Αλλά όχι όπω να είναι. Πρέπει να μπορούν να βρουν εργασία που να ε, είναι σε τομείς ποιότητας με σωστές συνθήκες εργασίας και με επαγγέλματα που σχετίζονται και με τις νέες τεχνολογίες. Εκεί όπου η αμοιβή είναι διπλάσια από τη μέση αμοιβή στις χώρες της Βαλτικής. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, θα τα πω αγγλικά Ε, διότι μου είναι πιο απλό. Αυτό που ακούσαμε από τον κ. Σικόσκι είναι ότι έχει ανησυχίες για το αν η Ευρώπη ακολουθεί το μοντέλο που είχαν φανταστεί οι ιδρυτές της το, την εποχή του κ. Άντενάουερ ή αν έχουμε παρεκτραπεί. Έχει αλλάξει πολύ η Ευρώπη έκτοτε. Έχουμε να κάνουμε μια τελείως διαφορετική Ευρώπη και ερχόμαστε και αντιμέτωποι με διαφορετική θέση των γυναικών στην οικονομία. Είναι διαφορετικές οι φιλοδοξίες του σήμερα και θα ήθελαν να συνδυάζουν τον επαγγελματικό και οικογενειακό βίο. Πρέπει λοιπόν να το αποδεχτούμε. Αυτό είναι ζωτική σημασία για τις στρατηγικές που αναφέραμε προηγουμένως. Εάν θέλουμε να χτίσουμε μια νέα Ευρώπη, μια ευφυή και αντιγωνιστική Ευρώπη, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το δυναμικό των γυναικών. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, θα χάσουμε. Θα είμαστε οι χαμένοι και μάλιστα οι χαμένοι σε σχέση με τους ίδιους τους δικούς μας τους στόχους της Ευρώπης του 2020. Θα πρέπει λοιπόν να σημειώσουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι πια η ίδια όπως πριν από 40-50 χρόνια. Και ε, τα δημογραφικά στοιχεία μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι γυναίκες που δεν έχουν δουλειά δεν κάνουν παιδιά. Έχουμε πολύ καλές δημογραφικές μελέτες του ΩΣΑ, αλλά και από άλλες χώρες σε εθνικό επίπεδο και δείχνει, δείχνουν όλες ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 90 άλλαξαν οι τάσεις. Προηγουμένως οι γυναίκες είχαν μια απασχόληση που ονομαζόταν κάπως μαξιλαράκι τρόπον την Δηλαδή οι γυναίκες πολλές φορές όταν δεν είχαν πολύ καλή δουλειά παράταγαν την επαγγελματικό βίο για να κάνουν παιδιά. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι γυναίκες που δεν βρίσκουν δουλειά δεν κάνουν καν παιδιά. Και βλέπουμε περιπτώσεις χωρών όπως η Σουηδία και άλλες σκανδιναβικές χώρες, όπου όταν οι γυναίκες προσπαθούν, μάλλον οι χώρες οι ίδιες προσπαθούν να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους σε αυτή τη συλλογιστική. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και για τους άντρε και για τις γυναίκες, όχι μόνο για τους άντρε, Διότι τον καιρό του Αντενάουερ υπήρχε η ιδέα ότι ο άντρα πρέπει να έχει μια σίγουρη δουλειά, ενώ η γυναίκα θα του υποστηρίζει λύνοντα τα οικογενειακά ζητήματα στο σπίτι. Τώρα πρέπει να αλλάξουμε τις νοοτροπίες. Αυτό συζητάμε και αυτό ακριβώ προσπαθούν να κάνουν οι στατικικές τις οποίες εκπονούμε και με τις οποίες πειραματιζόμαστε στην περιοχή της Βαλτικής. Μιλάμε για μια διαφορετική πλέον προσέγγιση. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω πολύ σύντομα και το θέμα της επιχειρηματικότητας. Προφανώς πρόκειται για ένα πολύ δυναμικό μερίδιο της τάσης δημιουργίας θέσεων απασχόλησης παντού. Το να συμπεραίνουμε ότι οι γυναίκε επιχειρηματίε είναι ίδιε με του άντρε επιχειρηματίε δεν μα πάει πουθενά. Διότι πέραν του να είναι επιχειρηματίε οι γυναίκε, πρέπει να φροντίσουν και την οικογένεια και τα παιδιά. Και αυτό πραγματικά απορροφά πολύ από την επιχειρηματική του ε, ενέργεια, για να το πω έτσι. Πρέπει λοιπόν και αυτό να το σκεφτόμαστε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι οι γυναίκε είναι το ίδιο με του άντρε. Για παράδειγμα, στην Πολωνία, αν μια άνεργη γυναίκα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια μικρή εταιρεία, ε, ρισκάρει να μην λάβει επιδόματα, ούτε άδειε που είναι μέρος των οφειλμάτων ε, ανεργίας, διότι δεν είναι επιχειρηματίας. Εάν λοιπόν πρέπει να αναλάβει τον κίνδυνο να ξεκινήσει μια επιχείρηση, τι άλλο διακινδυνεύει ότι θα έχει χαμηλότερη προστασία από την κοινωνική πρόνοια. Είναι λοιπόν θέματα θεωρητικά ναι και είναι θέματα νοοτροπία. Αυτά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με τα προγράμματά μας και τη στρατηγική αυτή. Αυτά θέτουμε προ συζήτηση και έχουμε και εμπειρίε αποδείξει από την πράξη τα πρότυπα που προσπαθούμε να ε, προωθήσουμε, να πιέσουμε δηλαδή τις γυναίκες να μένουν σπίτι για να κάνουν παιδιά μέσω των κοινωνικών εφολεμάτων και των παραδοσιακών οικογενειακών πολιτικών, βλέπουμε ότι δεν δίνουν αποτελέσματα. Θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι τέτοιε πολιτικέ δεν λειτουργούν. Διότι δεν υπάρχει θετικό αντίκτυπο. Το βλέπουμε, το βλέπουμε ότι είναι δαπανηρέ, με συγχωρείτε, αλλά μιλάω πολωνικά γιατί παθιάστηκα. Ε, ήθελα να το σχολιάσω και στα πολωνικά. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε στις γυναίκες ε, τη δυνατότητα να έχουν ε, τα καλύτερα δυνατά ε, ωφέλη από το να κάνουν παιδιά, τελικά έχουμε οδηγηθεί σε αποτυχία. Δεν λειτουργούν αυτέ τι πολιτικέ. Η Δημοκρατία τη Τσεχία, η Πολωνία προσπάθησαν να ε, ελοπίσουν υλοποιήσουν τέτοιε πολιτικέ που δεν έδωσαν αποτελέσματα. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι ήρθε πια η στιγμή να αλλάξουμε, να αλλάξουμε την προσέγγιση μας, τον τρόπο που βλέπουμε αυτά τα θέματα. Να συμμετάσχουν πραγματικά οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Όχι με επιφανειακό ή τεχνητό τρόπο όμως. Δεν θέλουμε να πιέσουμε κανένα να κάνει τίποτε. Όμως πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Για τις μεταφορές λόγου χάρη. Δώσαμε το παράδειγμα των αυτοκινητοδρόμων. Προφανώς θα πρέπει και η ισότητα των φύλων να ληφθεί εδώ υπόψη με τρόπο πραγματιστικό και όχι θεωρητικό. Σκεφτείτε τις αστικές συγκοινωνίες τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχουν δύο διαφορετικά διαμερίσματα. Θα έπρεπε λοιπόν να το λάβουμε υπόψη και στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας και στις πόλεις και στις περιφέρειες. Μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε πραγματικά να μας ε, βοηθήσει να βελτιώσουμε τα πράγματα σε μακροπεριφερειακό επίπεδο. Πρέπει να συγκεντρώσουμε τις διαφορετικές εμπειρίες των διαφορετικών χωρών της Βαλτικής και να αντλήσουμε διδάγματα. Αυτό θα μας επιτρέψει να αναθεωρήσουμε τις τοπικές και εθνικές μας ταπτικικές στη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι μια από τις προτεραιότητές μας σε όλες τις περιφέρειες της Πολωνίας. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να ολοκληρώσουμε με το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και να περάσουμε στο επόμενο, το σημείο 10, παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια στρατηγική για την περιοχή της Αδριατικής θάλασσας και του Ιουνίου Πελάγους θα δούμε σε πώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα σε σχέση με την εκπόνηση αυτής της στρατηγικής. Έχετε το λόγο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Hello, thank you very much. Good afternoon everybody. Good evening. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Έχω μία παρουσίαση PowerPoint, σας υπόσχομαι ότι θα είναι σύντομη, με την οποία θα προσπαθήσω να κάνω μία επισκόπηση της ε, προετοιμασίας για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή της Εδερτικής Θάλασσας και του Ιωνίου Πελάγους. Θα σας πω πώς έχει η κατάσταση σήμερα, αυτή την περίοδο και ποια είναι τα μελλοντικά βήματα κατά την προετοιμασία της νέας αυτής στρατηγικής. βάση για αυτή τη νέα μακροπεριφερειακή στρατηγική Ιωνίου και Αντρατικής είναι πολλές διαφορετικές πρωτοβουλίες συνεργασίας στην περιοχή αυτή και θα αναφερθώ κυρίως στην πρωτοβουλία Αντρατικής Ιωνίου και τα σχετικά φόρα, τα οποία ξεκίνησαν από το 2000 από την Αλβανία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη Σλοβενία. Έχουν περάσει πάνω από 14 χρόνια λοιπόν από τότε. Ξεκινήσε η συνεργασία αυτή μέσω μιας πρωτοβουλίας για τη σταθεροποίηση της περιοχής μετά από μία περίοδο συγκρούσεων και εξελίχθηκε τελικά η συνεργασία αυτή σε μία διακυβερνητική πρωτοβουλία για την περιφερειακή, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Ως αποτέλεσμα λοιπόν της πρωτοβουλίας αυτής βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε μια θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο, την οποία προτίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2012 και βάσει της στρατηγικής αυτής το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2012 έδωσε εντολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υποβάλει μια νέα πρόταση ε, στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο μέχρι τα τέλη του 2014. Πέρα από την εντολή αυτή που δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπήρχε και μία κάποια προϋπόθεση, ουσιαστικά να αξιολογηθεί καταρχάς η όλη έννοια της μακροπεριφερειακής στρατηγικής, πράγμα το οποίο είχε ζητηθεί ήδη από το Συμβούλιο προς την Επιτροπή πριν το 2011, και ζητήθηκε τον Ιούνιο του 2013 να παρουσιαστεί η αξιολόγηση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πω γι' αυτό λοιπόν δύο λόγια, αν μου επιτρέπετε. Αναφέρομαι λοιπόν στην αξιολόγηση αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2013, όπου ουσιαστικά λέγεται ότι οποιαδήποτε νέα στρατηγική θα πρέπει πρώτον να λάβει χώρα μόνο πραγματικά υπάρχει ουσιαστική ανάγκη και αν επιφέρει μια προστιθέμενη αξία για την συνεργασία μεταξύ κρατών μελών ή τρίτων χωρών, αν προβλέπετε κάτι τέτοιο από τη γεωγραφική περιφέρεια την οποία μελετούμε και στην αξιολόγηση επίσης λεγόταν ότι θα πρέπει οποιαδήποτε νέα στρατηγική να έχει συγκεκριμένους στόχους, να αντιμετωπίζει κοινέ προκλήσεις και να ανταποκρίνεται σε κοινέ ευκαιρίες για την περιφέρεια αυτή. Αναφερόμαστε λοιπόν σε μια προστιθέμενη αξία και σε κοινέ προκλήσεις. Πέρα από αυτά στην αξιολόγηση λέγεται ότι οι στρατηγικές αυτές, μάλλον ότι οι κύριοι της στρατηγικής αυτής ε, είναι οι ίδιες οι χώρες, άρα πρέπει πέρα από την πολιτική δέσμευση οι χώρες αυτές να διασφαλίζουν ότι θα υπάρχει απαραίτητη ηγεσία και διοικητική υποστήριξη για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Εθνικές Αρχές των οκτών αυτών χωρών που εντάσσονται σε αυτή τη νέα μακροπεριφερειακή στρατηγική συζήτησαν και εντόπισαν τέσσερις βασικούς πυλώνες για περαιτέρω ανάπτυξη. Ποιοι είναι αυτοί οι πυλώνες τώρα. Οι πυλώνες, μάλλον αυτοί, οι πυλώνες με συγκεντρώνουν τις περισσότερες ευκαιρίες και προκλήσεις. Πρώτον, θαλάσσια και ναυτιλιακή ανάπτυξη, δυνατότητα σύνδεσης, ιδίως όσον αφορά την ενέργεια και τις μεταφορές, περιβάλλον και τουρισμός. Έχουμε και δύο οριζόντιους τομείς, δημιουργία ικανοτήτων, καθώς επίσης και έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να πούμε ότι η θαλάσσια στρατηγική η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο έχει ενσωματωθεί, καλύπτεται πλέον από τις ε, ευρύτερες αυτές θεματικές ενότητες που έχουμε στην ευρωπαϊκή αυτή μακροπεριφερειακή στρατηγική. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε και τον πρώτον πυλώνα, ο οποίος αναφέρεται στην θαλάσσια ναυτιλιακή στρατηγική. Βλέπετε και τους υπόλοιπου πυλώνε, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά του έχουν σωματωθεί και αναφέρομαι στην ενέργεια, τι μεταφορέ κτλ. Τώρα την περίοδο από το Σεπτέμβριο έως την προηγούμενη ουσιαστικά εβδομάδα Μία ευρεία διαβούλευση έγινε στις 8 αυτές χώρες. Οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες, οι ενδιαφερόμενοι φορείς συμμετείχαν σε διασκέψεις υπό το συντονισμό των ίδιων των χωρών που συμμετέχουν στρατηγικοί. στρατηγική. Είχαμε ουσιαστικά ζευγάρια χωρών, ένα κράτος μέλος και ένα μη κράτος μέλος Βλέπετε ότι στην αρχή όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα υπεύθυνε ήταν η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο, στη συνέχεια για τη συνδετικότητα Ιταλία και η Σερβία, για το περιβάλλον η Σλοβενία και η Βοσνία Ζεγοβίνη και τον τουρισμό η Κροατία και η Αλβανία. Επίση έγινε και μία online δημόσια διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Οκτώβριο στον Ιανουάριο. Πρέπει να σας πω ότι στι διαβουλεύσεις αυτές λάβαμε πάρα πολλέ παρατηρήσεις και από άλλα θεσμικά οργανά, από την Επιτροπή των Περιφερειών συγκεκριμένα. Ξέρετε ότι υπάρχει μια διαπεριφερειακή ομάδα που έχει δημιουργηθεί στην Επιτροπή των Περιφερειών, ειδικά για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος. Είχαμε επίσης, λοιπόν, είχαμε μια πολύ σημαντική συμβολή από αυτές τις διαπεριφερειακές ομάδες και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή μετά από δικό μας αίτημα αποδέχθηκε να υποβάλει μια διερευνητική γνωμοδότηση που θα ενσωματωθεί και αυτή στην προετοιμασία της στρατηγικής αυτής. Βλέπετε λοιπόν ότι είχαμε μια πολύ σημαντική συμμετοχή από διάφορα όργανα. Στη συνέχεια έκλεισε αυτή η περίοδος διαβούλευσης με μια πολύ σημαντική διάσκεψη ενδιαφερομένων που έλαβε χώρα στις 6 και 7 Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Εστέφθη με επιτυχία 900 περίπου άτομα καταχωρήθηκαν, εγγράφηκαν στη διάσκεψη αυτή, αλλά δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη αίθουσα και μόνο 650 μπόρεσαν να παρευρεθούν. Προέρχονταν από όλες αυτές τις ε, περιοχές ε, τη στρατηγικής. Ο Πρωθυπουργό Ελλάδας Αντώνης Σαμαράς ε, προσφώνησε τη διάσκεψη αυτή. Πολλοί υπουργοί Έλληνε επίση ήταν ε, παρόντες και πήραν το λόγο. Επίτροποι, η κυρία Διαμανάκη συγκεκριμένα ήταν παρόντες. Και ξέρετε, ο Επίτροπος Χάν επίση και ξέρετε ότι η στρατηγική αυτή υπάγεται στις αρμοδιότητες της Επιτρόπου για θαλάσσια θέματα εφόσον όπως σας είπα σωματώνεται τη θαλάσσια διάσταση, η θαλάσσια πολιτική στη στρατηγική αυτή. Ποια είναι τα βασικά μηνύματα τα οποία εστάλησαν από τη διάσκεψη αυτή προς ενδιαφερόμενα μέρη. Η στρατηγική αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να κινηθούμε περισσότερο στο μέλλον, να ξεφύγουμε από την κρίση, να σημειώσουμε πρόοδο και λέμε επίσης ότι τέσσερι από τις οχτώ χώρε στρατηγικές αυτή είναι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι υποψήφιες ή δυνάμει υποψήφιες χώρες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λέγεται λοιπόν ότι η στρατηγική αυτή θα μπορούσε να υποστηρίξει επίσης την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων. Στα επιμέρους σεμινάρια που έλαβαν χώρα συζητήσαμε συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής της δράσης και τους στόχους για κάθε ένα θεματικό πυλώνα που αποτελούν τμήμα της στρατηγικής. Τώρα, πώς έχουν τώρα τα πράγματα. Ολοκληρώθηκε αυτή η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εξελογούμε αυτή τη στιγμή όλες αυτές τις παρατηρήσεις που λάβαμε και το τελευταίο αυτό διάστημα από τη διάσκεψη αυτή στην Αθήνα και θα προχωρήσουμε τώρα στην ίδια την κατάρτιση της στρατηγικής όπου θα έχουμε συγκεκριμένα μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένα σχέδιο δράσης. Θέλουμε μια ουσιαστική, ρεαλιστική στρατηγική όπου θα εντοπίζονται συγκεκριμένες προκλήσεις και ευκαιρίες αυτές που συζητήσαμε συγκεκριμένα στην Αθήνα και θα έχουμε ένα περιορισμένο αριθμό δράσεων που θα επικεντρώνονται στο τομείς εκείνους από τους οποίους μπορεί να προκύψει προστιθέμενη αξία. Ο γενικότερος στόχος στρατηγικής είναι η πρόθεση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, η δημιουργική οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασία στην περιοχή της Αντριατικής και του Ιωνίου, αλλά ένας επιπρόσθετος στόχος στρατηγικής είναι να διαδραματεί η στρατηγική αυτή ένα σημαντικό ρόλο στην πρόθεση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων και κυρίως των τεσσάρων αυτών μη κρατών της Ευρωπαϊκής, ε, ε, μη, κρατών που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήσαμε επίσης και την καλάζια ανάπτυξη με τους stakeholders. Αναφερθήκαμε συγκεκριμένα σε τομείς όπως η αλληλεία, η δατοκαλλιέργεια, οι θαλάσσιες ναυτιλιακές υπηρεσίες. Στο δεύτερο πυλόν αναφερθήκαμε στην συνδεκτικότητα, αναφερθήκαμε σε ενεργειακά δίκτυα και δίκτυα μεταφορών. Οι θαλάσσιες μεταφορές βέβαια είναι πολύ σημαντικές για αυτή την περιοχή, αλλά και οι ε, εγχώριες επίσης μεταφορές και οι διατροπικές μεταφορές. Και αναφερθήκαμε επίσης και στα ενεργειακά δίκτυα και το πώς μπορούν τα δίκτυα των κρατών αυτών να συνδέονται με ένα κεντρικό ε, δίκτυο παροχής ε, ενέργειας. Είπαμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας αυτής. Ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με την περιβαλλοντική ποιότητα, με το θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αναφερθήκαμε και σε άλλους τομείς όπως η βιοπικιλότητα, καθώς επίσης και η διατήρηση των διαφόρων ε, διαιτημάτων. Ο τέταρτος πυλώνας έχει να κάνει με τον βιώσιμο τουρισμό. Παρουσιάστηκαν οι στόχοι του τομέα αυτού και στην Αθήνα και είπαμε, μας είπαν στη συνέχεια ότι θα έπρεπε να αλλάξει ενδεχομένω κάπως ο τίτλος του τομέα αυτού, να λέμε καλύτερη βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού. είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε και κάποιους οριζόντιους στόχους όπως η υποστήριξη της διοικητικής ικανότητας παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες στην περιοχή αυτή καθώς επίσης και η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τώρα ποια είναι τα μελλοντικά στάδια. Από τώρα μέχρι τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντάξει την ανακοίνωσή τη και το σχέδιο δράση, λαμβάνοντα υπόψη όλε τι παρατηρήσει που έχουν υποβληθεί και στόχο μα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει τη σχετική στρατηγική και ουσιαστικά αναφέρομαι στην ανακοίνωση και στο σχέδιο δράση στα μέσα περίπου του Ιουνίου του 2014. Στη συνέχεια η στρατηγική θα κατατεθεί επισήμως στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 24ης Ιουνίου υπό Ελληνική Προεδρία ήδη προβλέπει στην ημερήσια διάταξή του τη συζήτηση της ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα με τη στρατηγική αυτή θα ασχοληθεί η Ιταλική Προεδρία που περιμένουμε και την επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το φθινόπωρο του 2014 σύμφωνα με την εντολή που έχει ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να ολοκληρωθεί δηλαδή αυτή η στρατηγική μέχρι τα τέλη του 2014. Στη συνέχεια, μετά την έγκριση αυτή, θα ξεκινήσει και η επίσημη υλοποίηση της στρατηγικής. Τώρα, η τελευταία μου διαφάνεια και το τελευταίο μήνυμα που θέλω να δώσω, ξέρετε ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές δεν έχουν συγκεκριμένα κονδύλια, δεν προβλέπονται για αυτές συγκεκριμένα κονδύλια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμως τα απαραίτητα ταμεία, υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, Βρισκόμαστε στην αρχή της νέας περίοδου, επομένως οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο να ευθυγραμμίσουν κάπως τα ταμεία εκείνα τα οποία ανταποκρίνονται στους κοινούς αυτούς στόχους και τις κοινέ ευκαιρίες που έχουμε στις περιφέρειες αυτές. Μέσω λοιπόν των μακροπεριφερειακών αυτών στρατηγικών θα πρέπει να καταφέρουμε να συντονίσουμε καλύτερα τα μέσα χρηματοδότησης που έχουμε για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, Ευχαριστώ. Κύριε Χρυσόγελος, παρακαλώ. Ε, ήθελα να κάνω μερικέ ερωτήσει, μερικές ερωτήσεις, some questions about that. Ε, οι, οι πυλώνες, οι τέσσερις που αναφέρονται, πώς επικοινωνούν μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τα θέματα της ενέργειας, πώς αυτό είναι συμβατό με το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Γιατί μιλάμε μόνο για τα δίκτυα με φυσικό αέριο ή ε, πετρέλαιο ή ηλεκτρική σύνδεση ή μιλάμε για ανανόσιμες πηγές ενέργειας για ένα συνολικό σχέδιο για την ενέργεια. Όταν μιλάμε για τον τουρισμό πόσο συνδέεται με, το, με, με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Ε, μιλάμε για ένα καινούριο σχέδιο το οποίο θα βαστεί σε πιο αποτελεσματικά πλοία από άποψη ενέργειας ε, που θα χρησιμοποιούν ανανόσιμες πηγές περισσότερο ε, περιβαλλοντική διαχείριση των λιμανιών ή απλώς για κατασκευή λιμανιών. Γιατί όλα αυτά που συζητάμε πρέπει να συνδέονται με το γεγονός ότι θέλουμε να είναι πιο πράσινες οι επενδύσεις, τουλάχιστον από το Ταμείο Συνοχής και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που εμείς τουλάχιστον εδώ στην Επιτροπή προσπαθήσαμε να το κάνουμε λίγο πιο πράσινο. Φοβάμαι ότι, ε, επειδή έχω συμμετάσχει ως ορισμένε συζητήσει, ε, υπάρχει μια παλιά προσέγγιση όλα αυτά. Δηλαδή, περισσότερα λιμάνια να προσεγγίζουν μεγάλα κουρασγερόπλια. Αυτό όμως δεν συνδέεται με βιώσιμες μορφές τουρισμού. Επίσης, αυτό που στάγαμε μόλις πριν, το θέμα της ενσωμάτωσης, της πολιτικής φύλου και ισότητας, πώς το λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό, από τη στιγμή που γίνεται η συζήτηση σε επίπεδο βαλτικής, γιατί δεν αξιοποιείται η εμπειρία και στις άλλες μακροπεριφέρειες, όπως είναι παράδειγμα Ιωνίου και Ανδριατικής, που είναι μια καινούρια ε, μακροπεριφέρεια. Αλλά πώς αξιοποιείται αυτή η εμπειρία. Η Βαλτική, για παράδειγμα, επενδύει αυτή τη στιγμή σε ένα δίκτυο φυσικού υγροποιημένου αερίου, το LNG. Η περιοχή Ιωνίου και Αδριατικής θα επενδύσει σε ανανόσιμε μορφές ενέργειας, που είναι διαθέσιμες στην περιοχή. Ε, χρειάζονται ορισμένε τομέ, γιατί αλλιώ φοβάμαι ότι άλλα συζητάμε για την περιφερειακή ανάπτυξη, άλλα θα είναι οι προτεραιότητε στου κανονισμού ο σχεδιασμό όμω βασίζεται σε παλιέ προσεγγίσει. Έτσι, δηλαδή, και επίση πρέπει να υπάρχουν ορισμένα όρια. Δηλαδή, συνδέουμε μεταξύ του ποια λιμάνια. Δηλαδή, ε, θα κάνουμε βαριέ υποδομέ για να πηγαίνουν μεγάλα κρουαζιερόπλια μία-δύο φορέ, τρει φορέ το χρόνο. Ή θα συνδέσουμε μεταξύ του διαδρομέ και άλλε για τον τουρισμό. Δηλαδή, που βασίζονται σε εμπειρίε, σε γνώσει, σε οικολογικέ μορφέ τουρισμού. Μιλάμε για βαριέ υποδομέ ή μιλάμε για πιο πράσινες υποδομές. Ε, φοβάμαι ότι αυτή η συζήτηση είναι πολύ ε, οριακή στη συζήτηση με τις μακροπεριφέρειες, αν και εμείς και σαν ομάδα των πράσινων είχαμε στηρίξει τις μακροπεριφέρειες, αλλά νομίζω ότι η συζήτηση που γίνεται στα διάφορα φόρα είναι τουλάχιστον μιας 15 ετίας, 20 ετίας πριν. Και δεν έχει λάβει υπόψη ε, όλα όσα συζητάγαμε εν ώψη των ταμείων αυτών. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια. Θέλετε να απαντήσετε, παρακαλώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θα παρακαλέσω την παρακαθήμενη συνάδελφο που παρακολουθεί ιδιαίτερα τα θέματα του τουρισμού να με βοηθήσει στην απάντηση. Να πω δύο λόγια σε σχέση με αυτά που είπατε κύριε Χρυσόγελε. Είναι η τρίτη στρατηγική για μακροπεριφέρεια αυτή. Και έχουμε την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να βασιστούμε στην εμπειρία των άλλων δύο στρατηγικών. Και να είστε βέβαιος ότι αυτό ακριβώς πράττουμε. Προσπαθούμε να βασιστούμε ε, και στα διδάγματα που βγάλαμε και στα σφάλματα και στην εμπειρία από αυτές τις άλλες δύο στρατηγικές. Εστιάζουμε για να αρχίσουμε σε πολύ λίγα θέματα και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα διδάγματα που μάθαμε από τη στρατηγική της Βαλτικής για τις προτεραιότητες και τα θέματα ε, που ήταν ευρύτατα όπως γνωρίζετε χωρίς αμφιβολία και για το Δούναβι. Λοιπόν, έχουμε περιορίσει τα θέματα, βασιζόμαστε σίγουρα στην εμπειρία μας και για τη διάρθρωση και τη δομή και για το περιεχόμενο της στρατηγικής. Αναφερθήκατε στο θέμα της ενέργειας η αηφορία και η βιωσιμότητα. Εγώ δεν το ανέφερα αυτό ως οριζόντιο θέμα η εγκάρσιο, διότι είναι προφανές ε, βεβαίω και θα πρέπει να προσπαθούμε ε, ενδεχομένω να το καθιστούμε πιο ορατό, να το προβάλλουμε περισσότερο. Αυτή η στρατηγική προωθεί ένα βιώσιμο και αηφόρο τουρισμό με ένα πυλώνα το περιβάλλον και την ποιότητά του. Όταν συζητούμε με τις εθνικές αρχές και τους ενδιαφερομένους και τους παίκτες εκεί, αυτό κάνουμε, ε, είναι αποτέλεσμα πολύ περιστατωμένη συζήτηση με τους ενεχομένους. Το ένα βασικό ήταν ότι ό,τι μπορεί να γίνει σε πιο αποτελεσματικό τρόπο και σε εθνικό επίπεδο ε, να συνεχίζεται να γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Η προστιθέμενη αξία και αυτή είναι άλλη μια έννοια κλειδί ε, εκτός από την αισίαση, θα πρέπει να είναι ακριβώς στο να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις ή ακόμα και ευκαιρίες που μπορούν να γίνουν καλύτερα σε συνεργασία ε, με τις χώρες. Για την ενέργεια, επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα ιδιαίτερο παράδειγμα. Ε, τουλάχιστον στην αρχή επιλέξαμε να εστιάσουμε σε δίκτυα, στη διασύνδεση ε, των διαφόρων grid μεταξύ των διαφόρων περιοχών, διασυνοριακά δηλαδή. Η πράσινη ενέργεια, εγώ δεν είμαι ειδικό στην πράσινη ενέργεια, επαναλαμβάνω ε, όσα μαθαίνω από τους ειδικού στις διάφορες χώρες, ε, έχει να κάνει με το εξής. Οι εναλλακτικέ πηγές ενέργειας είναι ανεπτυγμένες σε κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά χρειάζεται διασύνδεση των δικτύων, των grids μεταξύ των κρατών μελών για να κυκλοφορεί αυτή η ενέργεια και να μπορεί να αποδώσει. Και ε, αυτό έχω μάθει από τις συζητήσεις. Και τώρα εκεί μας ενδιαφέρει η διασύνδεση κυρίως του ηλεκτρικού δικτύου αλλά και η αγωγή. Για τον τουρισμό. Στόχος μας δεν είναι να φτιάξουμε νέες υποδομές μεγάλες. Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι και θα είναι να χρησιμοποιήσουμε την υφιστάμενη υποδομή με καλύτερο τρόπο με συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των κρατών της περιοχής έτσι ώστε να υπάρχει ε, αξιοποίηση και καλύτερο σχεδιασμό των νέων υποδομών σε περίπτωση που χρειάζονται. Και ιδιαίτερα για τον τουρισμό η βασική εστίαση είναι η βελτίωση της ποιότητας, διαχείριση του τουρισμού ακριβώς σε συνεργασία μεταξύ των κρατών στην περιφέρεια και προσβασιμότητα, δηλαδή να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει αρκετό συντονισμός μεταξύ των κρατών έτσι ώστε η προσφορά η τουριστική να είναι προσβάσιμη σε ενδεχόμενες αγορές. Νομίζω αυτά μπορώ να σας πω. Θέλω να δώσω το λόγο, μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, στη συνάδελφό μου για να συμπληρώσει μερικά πράγματα για τον τουρισμό. Να είστε βέβαιος ότι η πρόθεσή μας δεν είναι να έχουμε παλιωμοδίτικο σχεδιασμό ούτε από πάνω προς τα κάτω. Το αντίθετο, η μακροπεριφερειακή στρατηγική είναι κάτι που ζήτησαν οι χώρες. Δεν το επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τη βάση προς την κορυφή ήρθε αυτό το αίτημα. Και πάρα πολύ στεναρά ε, παρακάλεσαν, έκαναν έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους βοηθήσει να προετοιμάσουν αυτή τη στρατηγική. Εμείς ακούμε όσο γίνεται περισσότερους ενδιαφερμένους και μια πλειάδα μάλιστα η μεγάλη ποικιλία και τους τελευταίους μήνες και στην Αθήνα και προσπαθούμε ε, να ε, έχουμε βάσει της εμπειρίας από τις άλλες δύο περιφέρειες ε, την καινοτομία που χρειάζεται. Δεν ξέρω, έχεις να προσθέσεις τίποτα για τον τουρισμό. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Actually, that what... Um, Στα αγγλικά. Αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι ότι είμαστε στη στενή συνεργασία με τις άλλες γενικές διευθύνσεις, ιδιαίτερα του περιβάλλοντος, σε όλους τους πυλώνες. Σημειώνουμε τη θέση των άλλων γενικών διευθύνσεων και επίσης και την πρώτερη εμπειρία των άλλων μακροπεριφερειών και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε παντού ε, πράσινη ανάπτυξη και φιλική προς τον, στο περιβάλλον. Αυτό δεν αναφέρατε. Πραγματικά εγγραφόμαστε σε αυτό το πλαίσιο όσο μπορούμε. Και για τον τουρισμό δεν θέλουμε μεγάλες υποδομές, ε, τεράστια κατασκευάσματα. Ε, θέλουμε αηφόρο βιώσιμο τουρισμό με συγκεκριμένες δράσεις και ε, φιλικές προς το περιβάλλον. Okay, thank you very much. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε αυτό το θέμα. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Θέλω να σας ενημερώσω ότι για τους συντονιστές τα σημεία που είναι στην ημερήσια διάταξη θα διεκπαιρεθούν γραπτός, οπότε δεν χρειάζεται να συνεδριάσουν οι συντονιστές, δεν έχω διάφορα να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα είναι μόνο ημερή Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. Είναι μια πάρα πολύ σύντομη, πλην ε, κρίσιμη ε, συνεδρίαση γιατί θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 24 Φλεβάρι στο Στρασβούργο. Λήξη συνεδρίασης. Ευχαριστώ.